Um, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών. Θέλω να καλωσορίσω θερμότατα κυρίως όλα τα νέα μέλη. Να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης πρώτα λοιπόν. Η κυρία Σοφίνετ Βέλτε ένα διαδικαστικό. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος όλων των Ολλανδών συναδέλφων αλλά και άλλων εθνικοτήτων. Θα σας παρακαλούσα να αποτίσουμε ένα φόρο τιμή στην αρχή της συνεδρίασης ε, στα θύματα του αεροπλάνου που κατερρύφθη την περασμένη εβδομάδα γιατί η επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε να το πράξουμε αυτό θα είναι μόλις το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια και νομίζω ότι είναι πολύ καιρό και θέλω να πω για τα πρακτικά ότι... να το πω... Έχω εκπλαγεί δυσάρεστα τουλάχιστον ε, από τη σιωπή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένου και του Κοινοβουλίου. Ούτε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου δεν αναφέρεται το γεγονός. Θα ήλπιζα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου να καλέσει αύριο το απόγευμα, να συγκαλέσει μάλλον ανοιχτή δημόσια διάσκεψη των Προέδρων για να συζητηθεί το θέμα και να μην περιμένει μέχρι το Σεπτέμβριο. Αλλά εκείνο που είναι πρόεδρο, εγώ δεν είμαι, τουλάχιστον η Λίμπε να αξιοποιήσει την ευκαιρία να δώσει ένα μήνυμα προ τον κόσμο. Ευχαριστώ Σοφή που το θέτεις. Ναι και για τα νέα μέλη. Να πούμε ότι επειδή δεν συνεδριάζει η Ολομέλεια, ε, τούτη εδώ η ίσως είναι το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό σώμα που βρίσκεται ακόμα σε συνεδρίαση. Πραγματικά να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων αυτών. very much. Σας ευχαριστώ πολύ. And thank you for raising the point, Sophie. Um, ευχαριστώ πολύ, Σοφή. So, colleagues, um, welcome to this. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ξέρω ότι είναι τώρα προς τα τέλη της ε, κοινοβουλευτικής ε, περίοδου και ανυπομονείτε όλοι να πάτε διακοπές. Έχουμε θέματα όμως και πολλά και σήμερα και αύριο ανακοινώσει του Προέδρου και πάλι για τους νέους βουλευτές θα ήθελα να εξηγήσω μερικά πράγματα. Όταν πρώτο ήρθα εγώ σε τούτη εδώ την Επιτροπή δεν μου εξήγησαν τίποτα. Μπορεί να είναι λοιπόν βαρετό αυτό που θα πω και ανιαρό για τους παλιούς αλλά για τους καινούριου χρήσιμο. Ε, στην αρχή κάθε συνεδρίασης έχουμε τις ανακοινώσεις του Προέδρου, είναι διάφορα ε, διαδικαστικά και ε, διατυπώς πρακτικά ζητήματα εγώ έλαβα και αυτό τον κατάλογο, το λαμβάνετε κι εσείς ε, ένα ε, πάκο για οδηγίες προς ναυτιλωμένους νέους βουλευτές. Εγώ δεν το διάβασα και κακώς έκανα. Ε, παρακαλώ να το διαβάσετε και παλιοί βουλευτές που ήσασταν σε άλλες επιτροπές. Είμαστε από τις μεγαλύτερες επιτροπές της συναπόφαση με τεράστιο φάσμα θεμάτων. Η γραμματεία μας έχει ετοιμάσει λοιπόν αυτό και το φάκελο. Παρακαλώ να το διαβάσετε, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο το έγγραφο ε, και καλύπτει διάφορα θέματα, είπαμε, αλλά εκτός αυτού έχουμε πλήρη επίγνωση εδώ στην Επιτροπή μας ότι ασχολούμαστε με θέματα που απαιτούν και κάτι άλλο. Και τώρα προσπαθούμε κάπως να χαρτογραφήσουμε τα πράγματα για τους συναδέλφους για να υποφεληθούν από την εμπειρία των παλαιότερων και οι νέοι αλλά και τα νέα μέλη της Επιτροπής μας. Γύρω στο φθινόπωρο θα γίνει αυτή η άσκηση λοιπόν χαρτογράφησης και θα καλύπτει κάποια ειδικά θέματα, αστυνομικά, άσυλο, δεδομένα, τράφικινγκ. Ε, ε, είναι μια σύνοψη των όσων ε, θα μας απασχολήσουν και με χρονολογική σειρά. Επίσης θα χαρτογραφηθεί το σύνολο της νομοθεσίας και της δουλειάς που μας περιμένει. Ε, και αυτά που έχουμε κάνει με τη σειρά, όλα ε, τα νομοθετικά κείμενα, η νομοθεσία, τα ψηφίσματα, οι γνωμοδοτήσεις, οι εκθέσεις και τα ονόματα των συναδέλφων. Δεν υπάρχει ένα σημείο που μπορείτε όλα αυτά να τα βρείτε συγκεκριμένα. Και αυτό είναι χρήσιμο πλέον όταν παρακολουθείτε μια έκθεση, όταν είστε σκιώδεις, εισηγητές ή κάτι τέτοιο. Και σας είπα τον Οκτώβριο περίπου θα είναι στην ιστοσελίδα μια τέτοια χαρτογράφηση, έτσι την ονομάσαμε, μια άσκηση χαρτογράφησης για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και σημαντικό για την Επιτροπή μας, απλούστατα από το φόρτο και το αντικείμενο που καλύπτουμε. Παρακαλώ προς το παρόν διαβάστε αυτό το φάκελο. Ένα άλλο λοιπόν θέμα που θέλουμε να έχουμε θεματικές ε, ε, ενότητες για όλα τα μέλη ενημέρωση εάν ε, χρειάζεστε για την προστασία δεδομένων και άλλα θέματα που είναι πολύ περίπλοκα και σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Επιτροπής και άλλους ειδικού για επιμέρους πολιτικές ε, σε μικρές ομάδες βουλευτών ε, θα ενημερωνόμαστε πριν μπούμε στην ουσιαστική δουλειά γιατί ορισμένα από τα θέματα είναι αρκετά περίπλοκα, ας πούμε ασφάλεια και αστυνομία, προστασία δεδομένων. Για να δούμε ποια είναι η εμπειρία σας και τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό ήταν το τρίτο λοιπόν που ήθελα να αναφέρω. Και το επόμενο θέμα, αν πούμε τώρα αμέσω στην ουσία της συνεδρίασης, στις 10.30 θα καλωσορίσουμε δύο υπουργούς της Ιταλικής Προεδρίας, θα ακούσουμε πρώτα ε, όμως ε, τη συζήτηση για το γενικό προϋπολογισμό. Και ένα από τα νέα μέλη μας, ο κύριος Τόμας Τσεχόφσκι, είναι συντάκτης της νομοδότησης και θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση για το γενικό προϋπολογισμό. Πρώτα όμως θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά ε, τον συνάδελφο. Και στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής. Επιτροπή πρώτα. Τζο Μαράν, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που δίνετε στην Επιτροπή το λόγο. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ όλου, να σας συγχαρώ για την, για την εκλογή σας στην Προεδρία της Επιτροπής. Εμείς ως Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προσβλέπουμε ε, στη συνεργασία μας μαζί σας. Θα ήθελα επίσης ε, να συγχαρώ τον κύριο Γιαμασκόφσκι, με συγχωρείτε για τον τρόπο που προφέρω το όνομά του, για την επιλογή του ως Γενικού Εισηγητή του Προϋπολογισμού. Το εύχομαι κάθε επιτυχία. Τέλος, θέλω να ε, καλωσορίσω στην Επιτροπή και πάλι κάποια από τα παλαιά μέλη της που επανεξελέγησαν και θα ήθελα να τους ευχηθώ bienvenue. Ε, περνάμε τώρα στο θέμα του σχεδίου προϋπολογισμού του 2015. Ευθύς εξ αρχής κάποια γενικά ζητήματα και να αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο συντάχθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχήν, το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το λεγόμενο MFF, ε, συντάχθηκε το 2014 και αποτελεί την σταθερή βάση επί της οποίας θα συνταχθούν όλοι οι προεβολισμοί μέχρι το 2012. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι οι πιστώσεις ε, για το 2015 για τα ταμεία και τα προγράμματα στους τομείς πολιτικής που αφορούν την Επιτροπή σας ε, αντιστοιχούν επακριβώς στα στοιχεία που προβλέπει το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα, το MFFF. Το, ε, το αίτημα για πιστώσεις πληρωμών έχει υπολογιστεί προσεκτικά που αντικατοτρεύει, αντιπροσωπεύει το ποσό για το ξεκίνημα των προγραμμάτων και το κλείσιμο των υφισταμένων. Όσον αφορά τους αποκεντραμένους οργανισμούς που είναι πάρα πολύ σημαντικοί στο δικό μας χώρο, δεδομένου ότι αποτελούν τον χώρο που γίνονται πολλά πράγματα, ο χώρος αυτά τα οποία έχουν ζητηθεί στηρίζονται στον προπολογισμό για τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για το διάστημα 2014-2020 που εγκρίθηκε πέρυσι τον Ιούλιο. Παρά τα αυτά, στην σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε υπόψη της το αποτέλεσμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ε, για φέτος το 2014. Φέρει πίν. Η Europol πήρε δύο επιπλέον θέσεις σε αυτή τη διαδικασία συνδιαλλαγής που θα παραμείνουν στον οργανισμό το σχέδιο προπολογισμού του 2015 συνεχίζουμε την πολιτική του να χρησιμοποιούμε τα ε, πλεονάσματα των προηγουμένων ετών, στην περίπτωσή μας του 2013, σε σχέση με, την 2000, με τη ε, συνεισφορά του 2015 στους οργανισμούς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή περιλαμβάνονται μόνο τα νέα κονδύλια που απαιτούνται για την εξασφάλιση σταθερότητας το 2015. Επιπλέον και σύμφωνα με τις διατάξεις του MFF για τους οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τιμωρήσει τους οργανισμούς που δεν χρησιμοποίησαν πλήρως τα κονδύλια που τέθηκαν πέρυσι στη διάθεσή τους. Με βάση αυτά έχουν επιβληθεί οι εξής ποινές. 2% μείωση για υποεκτέλεση των πιστώσεων ε, πάνω από 5% που ε, στον ΙΑΖΟ και 2% μίεση για την ακύρωση των πιστώσεων πληρωμών πάνω το 5% δηλαδή για τη μη χρησιμοποίηση πάνω του 5% του προϋπολογισμού που ήταν στη διάθεσή τους στο EU Lisa. Για να κλείσω τη σύντομη παρουσίασή μου θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία του 2015 και να τα συγκρίνω με τα φετινά του 2014. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό. 2015 σχέδιο προπολογισμού για την, για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το, νέο ταμείο, περιλαμβανομένου και της, περιλαμβανομένης και των, της του, Ταμείου Επιστροφής, έχει αύξηση 3% και 140% σε πιστώσεις πληρωμών. 2015 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων αύξηση σχεδόν 3% σε δεσμεύσεις και πάνω από 20% σε πιστώσεις πληρωμών. Και τα δύο είναι, αποτελούν σημαντικές αυξήσεις που θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε στις υφιστάμενες συμβατικές μας υποχρεώσεις. Αυτό είναι μια σωστή κρίση του Κοινοβουλίου πέρυσι σε σχέση με το 2013, ότι δεν ήταν επαρκής οι πιστώσεις πληρωμών ώστε να μπορέσουν να, πληρωθούν οι υποχρεώσεις που ήδη είχαν αναλάβει τα ταμεία. Αύξηση λοιπόν κατά 140% στον ένα χώρο και 22% στον άλλον, κατά τον ίδιο τρόπο. Σχέδιο προπολογισμού του 2015 για το πρόγραμμα δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης και των παλιών προγραμμάτων για την ναρκωτικ... πρόληψη των ναρκωτικών και τη δικαιοσύνη, 5% για τις δεσμεύσεις και 24% περίπου σε πιστώσεις πληρωμών. Τώρα, οι οργανισμοί από κοινού συνολικά είχε ετηθεί για τους έξι οργανισμούς στο τομέα των εσωτερικών το 2015 από την Κομισιόν αύξηση κατά πάνω από 10% σε σχέση με το 2014. Αυτή η σημαντική αύξηση προκύπτει κυρίως από δύο οργανισμούς, τη Europol που ε, ε, παίρνει αύξηση 13% και η Ιουλίσα που είναι υπεύθυνη για το SIS και το VIS, θα είναι συστήματα πληροφορικής, κατά 22%. Το συνολικό, η συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τρεις αποκεντρωμένους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης το 2015 έχει μια μικρή αύξηση, λίγο πάνω από το 1% σε σχέση με το 2014. Ελπίζω ότι αυτή η γενική παρουσίαση θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε καλύτερα την πρόταση της Επιτροπής και να διευκολύνει τη συζήτησή σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, εισηγητή, τον κύριο Στυγκετόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα σύντομα ε, να ε, κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόταση αυτή. Τη διάβασα, την πρόταση Ευρωπαίκη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχω βασίσει και τη, ε, όλη μου προσπάθεια σε επιστολές που λάβαμε το Μάρτιο που απίφθηνανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον η δική μας Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζαμε τις επικρίσεις μας. Αν θέλουμε να αυξήσουμε τη ε, την χρηματοδότηση της Europol, Eurolis, ε, και Frontex και άλλων οργανισμών ε, που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην εσωτερική ασφάλεια. Δηλαδή, ε, τι εννοώ με όλα αυτά. Ότι είναι σημαντικό να αναλάβουμε ουσιαστική δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αυξήσει τον προϋπολογισμό των οργανισμών αυτών. Αυτό θα αυξήσει τελικά, πιστεύω, την ασφάλεια των πολιτών στην Ευρώπη. Κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι το εξής. Υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, και κάποια σημεία που πρέπει να σχολιάσουμε. Ας πούμε, προθεσμίες. Στις 27 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για τη γνωμοδότησή μας. Και στη συνέχεια, 1η ή 2 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε μια συνεδρίαση σε επίπεδο σκιωδών εισηγητών, ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ. Αυτά. Thank you very much. I think... Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι 27 ε, Οκτωβρίου είναι όντως η ε, ημερομηνία, ε, Αυγούστου, συγγνώμη, 27 Οκτωβρίου, ε, και θα το κοιτάξουμε και θα το ελέγξουμε ξανά. Ε, κάτι για τα νέα μέλη πάλι. Μάλλον κάποιος από τα νέα μέλη έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Φέσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω ως κοιόδης εισηγητής εκ μέρους της Άλντε. Αν είναι κατάλληλη στιγμή βέβαια είναι από ό,τι φαίνεται. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Άλντε υποστηρίζει τη γνωμοδότηση αυτή και συμφωνεί με τις προτεραιότητες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Τώρα περισσότερο παρά ποτέ είναι σημαντικό να υπάρξει ε, σοφροσύνη στη διαχείριση του προϋπολογισμού αλλά και επαρκή κονδύλια για να λειτουργήσουν οι οργανισμοί. Γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω αύξηση στον προϋπολογισμό της Frontex και θα παρακολουθούμε στενά τον στη σωστή χρήση των πόρων από τον οργανισμό. Θέλουμε να αυξηθεί το προπολογισμό ώστε να μπορέσει να είναι αποτελεσματική στα καθήκοντά της. Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν επαρκείς πόροι για τους άλλους ε, οργανισμούς που ε, συμμετέχουν στην ειδική ομάδα Μεσόγειος. Τώρα, ε, θέλουμε να υπάρχει περισσότερη διαθέσιμη πόρη στο θέμα του ασύλου και ίσως με μείωση του προπολογισμού σε, άλλους, σε άλλα κονδύλια. Στο πριν του τέλος ε, της προηγούμενης θητείας η Λίμπε ζήτησε την δικαιολόγηση της αύξησης του προπολογισμού του ίδιου e Λίζα. Τα μεγάλα συστήματα πληροφορικής δεν σημαίνουν κατά ανάγκη μεγάλες αυξήσεις του προπολογισμού. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε από την Επιτροπή να μας εξηγήσει σήμερα γιατί χρειάζεται αυτή η μεγάλη αύξηση. Και όσον αφορά στην τήρηση του νόμου θα πρέπει να δίνουμε εμείς το παράδειγμα. Στην ε, απόφαση της 8ης ε, Απριλίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, ε, ακύρωσε την ε, οδηγία για την διατήρηση δεδομένων. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε ακόμα εκτιμήσει πλήρως τις συνέπειες αυτής της απόφασης. Λοιπόν, θα μπορούσε η Κομισιόν να μας πει ε, ποιες, τι χρηματοδοτούν αυτές οι ε, καταστάσεις. Πριν να γίνει μια ενδελεχής νομική αξιολόγηση με σκοπό να, να, να συζητηθεί τι θα γίνει στην Κομισιόν σε σχέση με την διατήρηση των δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Δίας Δεμέρα, παρακαλώ. Κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο ε, πάρα πολύ εμπεριστατωμένο και σε μεγάλες λεπτομέρειες για τους ε, οργανισμούς αυτούς και θα ήταν μάλιστα και επικριτικά τα σχόλιά μου. Για ποιο λόγο. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι περισσότερες δαπάνες, αλλά να πιάνουν τόπο τα χρήματα και να εκτελούνται οι προϋπολογισμοί, να εκτελείται ο προϋπολογισμός στην κυριολεξία. Ε, για την Ευρωπόλ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Τι γίνεται εκεί. Ο προϋπολογισμός του 14 ήταν 88,6 εκατομμύρια, για το 15 προτείνεται 92,7 εκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία μου αυτό συνιστά αύξηση 12%. Η Κομισιόν το υπολογίζει 13%. Η αύξηση αυτή του προϋπολογισμού για την Ευρωπόλ ε, θα ε, πήγαινε σε δύο τομείς ουσιαστικά. Τα λειτουργικά συστήματα πληροφορικής και ε, η καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο. Με το προσωπικό μας τι γίνεται. Όπως γνωρίζετε μετά τη διοργανική συμφωνία για τον προπολογισμό του 2014 με 2020 είχαμε βάλει στόχο τη μείωση κατά 5% των υπαλλήλων στις 32 αυτές ε, υπηρεσίες οργανισμού οργανισμούς της Ένωσης κατά την επόμενη πενταετία. Στην πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μείωση ε, στο προσωπικό δύο συν να αυξηθεί με τέσσερις ε, συμβασιούχους ορισμένου χρόνου για το έργο των ε, προγραμμάτων πληροφορικής. Έτσι όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπόλ και να ανταποκριθεί στο έργο της. Είναι κατάφορη αυτή η αντίφαση και πολύ μεγάλη. Τι ζητάει η Ευρωπόλ, δεν ζητάει περισσότερα χρήματα. Γιατί τις έχουν δοθεί. Αλλά αυτό που θέλει η Ευρωπόλ θέλει ενίσχυση στο προσωπικό. Γιατί είναι αυξημένη η ζήτηση ε, των υπηρεσιών. Ζητάει 29 θέσεις συμβασιούχου για το EC3 και 10 για το EC3. Τι σημαίνει αυτό ότι χρειάζεται 3 εκατομμύρια ευρώ για μισθοδοσία αυτών των ε, συμβασιούχων. Προτείνει κάτι ο Τόμας, ο συντάκτης της γνωμοδότησής μας, τον οποίον επιφύλακτα υποστηρίζω και θα κάνω και μια τροπολογία που δεν είχα χρόνο ακόμα να υποβάλω και έχει ως εξής. Να είναι αυτές οι θέσεις ε, προσωρινές έκτακτων υπαλλήλων ε, συμβασιούχων. Και να πω και κάτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα. Άλλη κατάφορη, κατάφορη ε, πραγματικά αντίφαση από πλευράς της Κομισιόν. Όταν θέλησε να ε, συγχωνευθούν η ΣΕΠΟΛ και η Europol και δόξα το Θεό το Κοινοβούλιο αυτό το απέτρεψε, ε, μας έλεγε η Επιτροπή τότε και ισχυριζόταν ότι αν συγχωνευθούν θα είχαμε 17,2 ευρώ εκατομμύρια οι οικονομίες στην περίοδο 15 με 20. Παρ' όλα αυτά, για μία μόνο άσκηση, για ένα οικονομικό έτος μας ζητούν αύξηση κατά 12%. Και θέλω να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί πολύ προσεκτικά και αναλύει όχι μόνο την πρικοδότηση αλλά και την εκτέλεση στη συνέχεια του προϋπολογισμού με τα επιχειρήματα που προβάλλεται. Λοιπόν, Τόμας, εμείς θα υποστηρίξουμε τη γνωμοδότησή σου, θα κάνουμε αυτέ τι τροπολογίε αυτά τα ολίγα πρόεδρε και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Νίτα Μιουλάρ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Στεχόφσκι για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει σε τόσο σύντομο χρόνο και είναι και νέος βουλευτής. Γενικά πιστεύω ότι με βρίσκει σύμφωνο η γνωμοδότηση. Είναι, πιστεύω, αποτέλεσμα καλής ανάλυσης της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προπολογισμό του 2015. Έχω όμως πολύ συγκεκριμένες ανησυχίες και πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 3 που αφορά τις, τους ανεπαρκείς πόρους, της Γιουλίζα πιστεύω ότι υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων θα πρέπει να έχουμε πιο έντονη διατύπωση. Το πακέτο για το άσυλο που εγκρίθηκε το 2013 θα πρέπει να υλοποιηθεί τα επόμενα έτη να εκτελεστεί και αυτό σημαίνει επιπλέον ε, διοικητικό φόρτο και δεν μπορεί να μειώνεται ε, ο προϋπολογισμός ενός οργανισμού του οποίου τα επόμενα έτη θα πολλαπλασιαστεί η δουλειά. Θα κάνω αργότερα τροπολογία για την παράγραφο 3 αυτή. Εκτός αυτού, λοιπόν, θα πρέπει να πω ότι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράφες ανησυχούν γιατί στο σχέδιο προϋπολογισμού ε, της Ένωσης, τις εσωτερικές υποθέσεις, στον τίτλο 18, έχουν ε, προσημειώσει ε, περισσότερα κονδύλια για την, τον ε, επαναπατρισμό και επαναπροώθηση ε, των προσφύγων. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο συντονισμένη προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 5 και 6 πιστεύω ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ δεν θα πρέπει να καλωσορίσει καμία αύξηση σε τομεί που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαπραγματεύσει. Ο κανονισμός της Europol δεν έχει ακόμα εγκριθεί, ξέρετε. Οπότε οποιαδήποτε αύξηση του προϋπολογισμού της ε, ε, δεν ε, δικαιολογείται. Επιπλέον θα πρέπει να είμαστε και πιο ε, προσεκτική όταν μιλάμε για το πρόγραμμα εφηαιών συνόρων, για το σύστημα εισόδου και εξόδου. Είναι εξαιρετικά επίμαχο. Εγώ θα πρότεινα μια πιο προσεκτική διατύπωση. Γενικά, ναι, στη γνωμοδότηση και προβλέπω στη συνεδρίαση των σκιωδών. Ε, τελευταίο, χωρίς να είναι το λιγότερο αυτό σημαντικό, θα σας παρακαλούσα να ε, υποστηρίξετε την πρότασή μου για ένα πολιτικό Επιλωτικό συγγνώμη, πρόγραμμα με μοναδικό στόχο να υπάρχουν μεγαλύτερες συνέργειες ανάμεσα στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών και την περιφερειακή πολιτική αλλά και ε, τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να βελτιωθεί η εκπαίδευση των Ρωμά, ε, να εξαλειφθεί ο αποκλεισμός ε, και οι διακριτικές μεταχειρίσεις των παιδιών τους θα ενταχθούν καλύτερα οι Ρωμά ε, στην ε, Ένωση, αν είμαστε σοβαροί λέγοντας ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση και η εργασία για όλους είναι πραγματικός στόχος. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά τελευταία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα είμαι σύντομη, δεδομένου ότι δεν ε, έχω μελετήσει τα θέματα στις λεπτομέρειές τους. Όμως, είχα, ε, ε, μου έκανε κακή εντύπωση η ισορροπία του προεπολογισμού μεταξύ θεμάτων ασφάλειας και δικαιοσύνης αφετέρου και δικαιωμάτων των πολιτών. Οι μεγαλύτεροι προϋπολογισμοί είναι αυτοί που αφορούν τα λεγόμενα θέματα ασφάλειας, ε, όπου δεν υπάρχει ισορροπία για την, ισορροπία για την ασφάλεια, τα δικαιώματα και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το ίδιο ισχύει για τη Frontex όπως και για το άσυλο, τη μετανάστευση κλπ. Και συνεχίζω να μην είμαι ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο εξισορροπήθηκε το Ταμείο αυτό στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου του προπολογισμού έχουν αφαιθεί πάρα πολλά πράγματα στα κράτη-μέλη και βρισκόμαστε όλοι εδώ για να κάνουμε, να φροντίσουμε ότι, και το γνωρίζουμε, ότι στα κράτη-μέλη πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, ιδίως όσοι γνωρίζουμε το δράμα στη, της Μεσογείου. Θα κάνω προτάσεις τροπολογιών για του, στον εισηγητή και βεβαίως περιμένω ανυπόμονα τη συνειδρίαση των σκιωδών. Ε, χαίρομαι πολύ που την ε, ε, περιμένετε με ανυπομονησία. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι το πνεύμα μας. Θέλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε, βεβαίως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Όμως, τέθηκαν πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα στη διάρκεια των ομιλιών. Όλα τα σημειώσαμε σε σχέση με την Frontex EASO δύο θέματα. Πρώτον, τα ποσά που προβλέπει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2015 είναι αυτά που ζήτησαν οι ίδιοι οργανισμοί. Δηλαδή στηρίξαμε πλήρως τις προτάσεις των οργανισμών. Κατόπιν τούτου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο προϋπολογισμός δεν είναι οριστικός και μετάκλητος. Πρέπει να είναι και όντω είναι ένα ευέλικτο μέσο. Το γνωρίζετε γιατί συνεχώς ασχολείστε με την τροποποίηση των προπολογισμών. Αν αλλάξουν οι συνθήκες και όντω το δικό μας χώρο όντως αλλάζουν, πάντοτε υπάρχει δυνατότητα τροποποίηση των προϋπολογισμών και βεβαίως σε σχέση με τη Μεσόγειο όπου και η Frontex και ε, ο ΕΑΖΟ είναι πάρα πολύ δραστήριοι. Δεύτερον, ο Γενικός Διευθυντής μου κ. Χουτ θα έρθει να απευθυνθεί στην Επιτροπή σήμερα το απόγευμα για το θέμα της ειδική ομάδας Μεσόγειο και θα πρέπει να, να χρησιμοποιήσετε την ευκαιρία αυτή να συζητήσετε τα ζητήματα αυτά μαζί του. Ένα θέμα που ετέθη και το εκτιμούμε ιδιαίτερα είναι η ιδέα ότι δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να αυξηθεί ο προπολογισμό, αλλά να γίνονται καλύτερες δαπάνες. Πιστεύω ότι σε κάθε τομέα δαπανών υπάρχει περιθώριο να γίνουν περισσότερα με τα ίδια χρήματα ή να γίνουν περισσότερα και με λιγότερα χρήματα. Σημειώνω ότι τα θέματα της επάνδρωσης των οργανισμών είναι ένα ζήτημα που θέλουν οι βουλευτές να τεθεί και να το παρακολουθήσουμε. Το σημειώνουμε αυτό. Όμως έχουμε δεσμευθεί να μειωθεί το προσωπικό του, ε, των οργανισμών όπως συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να μειωθεί κατά 5%. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιτευχθεί. Όμως στο εσωτερικό των οργανισμών υπάρχουν μικρά περιθώρια ε, ελιγμών. Τέλος, σχετικά με αυτό που αναφέρθηκε για το EU και τη σημαντική αύξηση του προπολογισμού του. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση του ε, πληροφοριακού συστήματος Visa ε, που πρέπει να γίνει το 2015 και όσοι ασχολούνται με την πληροφορική γνωρίζουν ότι η σημαντική αναβάθμιση των μεγάλων πληροφορικών συστημάτων συνεπάγονται μεγάλο κόστος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να πω στους συναδέλφους ότι όπως και στο παρελθόν ε, προτείνεται να έχουμε μια προθεσμία υποβολής τροπολογιών 27 Αυγούστου, είναι η μέρα Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι και αυτό θα πρέπει να λάβετε υπόψη, θα πρέπει να γίνει μόνο στα αγγλικά. Είναι κρίμα, ε, ξέρω αν ε, έχετε ε, αντιρρήσεις, ελπίζω να μην έχετε, βεβαίως όμως μπορείτε να έχετε. Επίσης έχουμε εδώ τον κύριο Ντιπρέη που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής αλλά επίσης και πρώην ε, εισηγητής των προϋπολογισμών και ε, πρέπει να πω στους συναδέλφους ότι αν σας ακούγεται στεγνή αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή γιατί ασχολείται με, την, ε, το θέμα που επηρεάζει την ίδια τη λειτουργία και τη ζωή των οργανισμών. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και όπως έλεγε ο κύριος Ντυπρέ, ε, πρέπει, είναι, όλοι συμφωνούμε ότι είναι καλό αυτό. Επίσης όταν ανέλαβα την Προεδρία, ο πρώην ε, Πρόεδρος που δεν παρίσταται τώρα, ε, δεν ήταν εδώ. Οπότε με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας του θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα όσα προσέφερε στην Επιτροπή μας. Έχουμε λοιπόν δύο πρώην Προέδρους στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρώην Πρόεδρο, τον Φερνάντο. Δεν ξέρω αν τα καταλάβατε όλοι. Έχουμε δύο πρώην Προέδρους της Επιτροπής ε, Λίμπε μέσα στην αίθουσα, οι οποίοι όμως δεν ήταν εδώ όταν πρωτοανέλαβα εγώ. Έχω μια άλλη ανακοίνωση. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τα δανέζικα. Αν υπάρχουν δανείοι βουλευτές στην αίθουσα, μπορούν να μιλήσουν δανέζικα αλλά δεν μπορούν να ακούν τη γλώσσα τους. Ε, και από ό,τι βλέπω έχουμε τουλάχιστον έναν δανό. Ε, εξηγώ στα νέα μέλη ότι τέτοιου είδους ανακοινώσεις πρέπει να γίνονται, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να φροντίζουμε να έχετε διαρμηνία στις γλώσσες σας. Είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι ανακοινώσεις. Όπως βλέπετε έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, έχουμε ε, είμαστε τελειώσει νωρί τη συζήτηση. Κυρία Βερζέ, θέλετε να πάρετε το λόγο επί ποιου θέματος. Στο θέμα των ε, τροπολογιών, κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, πρέπει να κάνουμε τις τροπολογίες για τον προϋπολογισμό μόνο στα αγγλικά μέχρι τις 27 Αυγούστου. Και αν ξέρω να μετράω, είναι ένας μήνας και. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, αλλά προσπαθήσαμε στο παρελθόν, ακόμα και όταν μας πίεζαν πάρα πολύ οι ε, προθεσμίες, να αποφύγουμε τέτοιου είδους αδίέξοδα και ε, αδυναμία εργασίας στην, προσω... Ε, στη μητρική μας γλώσσα. Ας βάλουμε δύο προθεσμίες μια πιο σύντομη προθεσμία για τις τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες και μια πιο ευρύχωρη ας πούμε για τροπολογίες στα αγγλικά μέχρι και τελευταία στιγμή ας πούμε. Επειδή έχουμε και πολλά νέα μέλη, να μην αρχίσουμε τώρα με κακές συνήθειες με το καλημέρα σας, να δρομολογηθούν τα πράγματα σωστά με σεβασμό στην πολυγλωσία. um, I mean, we have... Κοιτάξτε, έχουμε ευελιξία να ορίσουμε τις 13 του μηνός για την κατάθεση τροπολογιών. Αν σας βοηθάει αυτό. Αν υπήρχαν αντιρρήσεις. Βεβαίως είναι και λογική και θεμητή. 13 λοιπόν του μηνός Αυγούστου αν συμφωνείτε. 13 Αυγούστου για να κάνετε τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες. Πάντα μεσημέρι είναι η προθεσμία, συνήθως στις 12 ε, λίγη. 13 Αυγούστου λοιπόν στις 12 το μεσημέρι και 3 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχω μια κατάσχετη φλιαρία, γιατί τελειώσαμε νωρίτερα. Για τα νέα μέλη, το λέω αυτό, στις 10.30 θα έρθουν οι υπουργοί. Ποιος θέλει το λόγο, παρακαλώ. Για αυτό το θέμα, για άλλο θέμα θέλεις. Μια στιγμή να τελειώσω αυτό. Λοιπόν, έλεγα στις 10.30 θα έρθουν οι υπουργοί από την Ιταλία να μας κάνουν τις προγραμματικές δηλώσεις. Ακόμα δεν έχουν φτάσει. Άννα, τι ήθελες να πεις εσύ, διαδικαστικό ήταν ή κάτι τελείως διαφορετικό. Γενικότερο. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Αρχίσαμε ε, τη συνεδρίαση με αυτό το θλιβερό γεγονός της κατάρριψης ε, του αεροσκάφους. Αλλά σας θυμίζω ότι πριν από τρία χρόνια 69 νέοι σοσιαλδημοκράτες στην Νορβηγία βρήκαν το θάνατο στην Ουτάγια και φτάσει στο Όσλο ε, στα κυβερνητικά κτίρια. Είναι σημαντικό να το θυμίσουμε και αυτό ως επέτειο, διότι κάποιος ήθελε να σκοτώσει κάποιους νέους που είχαν ελπίδες και πίστευαν στην κοινωνία, στην πολιτική ε, και ήταν ε, στρατευμένοι ε, σε αυτή την υπόθεση. Καλό είναι να μην το ξεχνούμε γιατί συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από αυτή την τραγωδία στην Νορβηγία. Ναι, το σημειώνουμε. Ας κάνουμε μια σύντομη διακοπή τώρα, ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να έρθουν οι Ιταλοί υπουργοί. Παρακαλώ μην απομακρυνθείτε πάρα πολύ, εδώ γύρω να μείνετε γιατί θα ξαναρχίσουμε αμέσως μόλις φτάσουν. Maybe. Colleagues, please take your seats. Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. colleagues, we're going to begin the meeting. Λοιπόν, συνάδελφοι, τη συνεδρίαση. Και πάλι μερικά τεχνικά πριν ε, αρχίσουμε και πρακτικά, πριν μπούμε στην Ιταλική Προεδρία. Για το προηγούμενο που συζητούσαμε για τον προπολογισμό, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 27 Αυγούστου. Το αποφασίσαμε έτσι τελικά και είμαι υποχρεωμένος να το ανακοινώσω εδώ από την έδρα για να είμαστε σύμφωνοι με τους κανόνες. Μπορώ να σας εξηγήσω εκτενέστατα και μέχρι ναυτίες, αλλά δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ε, με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε την ευκαιρία να υποδεχτώ δύο συναδέλφους της Ιταλικής Προεδρίας, τον Υπουργό Αλφάνο και τον Υπουργό Ορλάντο είχα την ευχαρίστηση και τη χαρά να εκπροσωπήσω το Κοινοβούλιο στο άτυπο Συμβούλιο Στερικών και Δικαιοσύνης και θα ήθελα να πω πριν ε, δώσω το λόγο και στους δύο υπουργούς ότι ήταν ε, εξαιρετικά καλή οργάνωση αυτού του Συμβουλίου με πάρα πολύ μεγάλη εστίαση, με οξύτητα στην Task Force και τη Μεσόγειο, στα θέματα μα στρατηγικές κατευθυντήρες γραμμές για την προστασία των δεδομένων, για το EPPO ήταν σχεδόν κατάλογος ε, των δικών μας προτεραιοτήτων ε, όλα τα θέματα του Συμβουλίου. Και για μας λοιπόν και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στράφηκε η συζήτηση σε θέματα που μας ενδιαφέρουν και μας ε, απασχολούν. Ε, Συρία, επανεγκατάσταση και βεβαίως και η πολιτική κατάσταση μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και πώς επηρεάζονται όλα αυτά τα ζητήματα. Πολύ καλή οργάνωση και σας ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα θα μάθουμε στη συνέχεια και θα έχετε όλο το χρόνο να κάνετε ερωτήσεις στους υπουργούς. Όπως είχα και εγώ την ευκαιρία στο άτυπο αυτό συμβούλιο. Λοιπόν, θα δώσω πρώτα το λόγο στον Υπουργό τον κύριο Αλφάνο για 10 λεπτά και μετά στον Υπουργό Δικαιοσύνης για 10 λεπτά στον κύριο Ορλάντο. Και θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Α, εξηγήσω στα νέα μέλη τι κάνουμε. Πρώτα, στον πρώτο γύρο μιλάνε οι συντονιστές. Εάν οι συντονιστέ στηρούν το χρόνο τους. Έχουμε απολύτως στη συνέχεια χρόνο να κάνουν ερωτήσεις στα υπόλοιπα μέλη. Ένα δεύτερο όμως γύρο ερωτήσεων. Ο κύριος Αντζελίνο Αλφάνο, Υπουργός Εσωτερικών, έχει το λόγο για ένα δεκάλεπτο το πολύ και αν τηρήσετε το χρόνο σας θα έχουμε χρόνο πολύ για ερωταπαντήσεις που θα είναι και πολλές ερωτήσεις με βέβαια. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μωράες, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε εδώ σήμερα στην Επιτροπή σας. Τον ευχαριστώ λοιπόν, διότι συμμετείχε επίσης και στην άτυπη συνεδρίαση που είχαμε στο Μιλάνο. Για μένα λοιπόν είναι ένα τεράστιο προνόμιο να βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα στη δική σας την Επιτροπή και στην αίθουσα αυτή η οποία είναι αφιερωμένη σε έναν πολύ μεγάλο Ιταλό πολιτικό ο οποίος πραγματικά έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σημαντικές αξίες ελευθερίας και ενοποίησης. Ένας άνθρωπος από τον οποίο, για τον οποίο μάλλον έχουν περάσει ή θα περάσουν μέσα σε μερικές εβδομάδες 60 χρόνια από το θάνατό του. Αναφέρομαι προφανώς τον Άλτσιντεν Ντεγκάσπερη. Γνωρίζω λοιπόν ότι ξεκινάει αυτή η Ιταλική Προεδρία, αυτό το εξάμεινο της Ιταλικής Προεδρίας, σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο μετάβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανανεώθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανανεώθηκε επίσης η, θα ανανεωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αρχίσει να λειτουργεί σύντομα μια νέα σύνθεση. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να πούμε εξ αρχής δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα να έχουμε μια καλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και πιστεύω ότι η δική σας Επιτροπή, από τη δική σας την Επιτροπή εξαρτώνται πάρα πολλά από τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα των δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της ασφάλειας είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, θεμελιώδης θα έλεγα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. συνεδριάζεται σήμερα ως Επιτροπή που πραγματικά διαχειρίζεται το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά έτσι βλέπω τα πράγματα. Εναπόκειται λοιπόν σε εσά και στο Συμβούλιο προφανώ να καταφέρουμε να έχουμε μια πλήρη συνεργασία. Στα πλαίσια τη συναπόφαση, ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικό, ουσιαστικό θα έλεγα, όχι μόνο για τα όσα απορρέουν νομικά από τη συναπόφαση, αλλά υπάρχει και μια έντονη πολιτική διάσταση είναι πολύ σημαντικός ο πολιτικός συμβολισμός της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της έγκρισης της κοινοτικής νομοθεσίας. Όσον αφορά τώρα τις εσωτερικές υποθέσεις, ποιες είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της Ιταλίας. Θέλουμε προφανώς να έχουμε για τις εσωτερικές υποθέσεις μια πολύ στενή σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να καταφέρουμε να προωθήσουμε τις πρωτοβουλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει και να προωθήσουμε και νέες πρωτοβουλίες και θα θέλουμε επίσης να προωθήσουμε και τις νέες κατευθυντήρες γραμμές τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει να επεξεργαζόμαστε και τις οποίες ήδη έχουν αναλύσει και οι υπόλοιπες, οι προηγούμενες προεδρίες και θα αναλύσουν και οι επόμενες προεδρίες, συγκεκριμένα προεδρία της Λετωνίας και, της, ε, του Λουξεμβούργου. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της μετανάστευσης, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό το οποίο καλούμεθα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε. Είναι η ιστορική στιγμή αυτή και πρέπει να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε ευρωπαϊκές απαντήσεις και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αφιερώσαμε μία συγκεκριμένη σύνοδο του Άτυπου Συμβουλίου του Μιλάνου που έλαβε χώρα στις 8 Ιουλίου. Με βάση λοιπόν τους στόχους της Task Force της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλάβουμε άμεση δράση προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε αποτελέσματα με άμεσες επιπτώσεις, αλλά χρειαζόμαστε επίσης και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις προκειμένου να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης. Να σας υπενθυμίσω ότι η δική ομάδα για τη Μεσόγειο δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο του Οκτωβρίου του 2013 μετά την ε, τραγωδία που είχαμε στα νυχτά της Λαπεντούζα όπου έχασαν τη ζωή τους 800 μετανάστες. Τότε ξεκίνησε, τότε συστάθηκε η δική ομάδα για τη Μεσόγειο. Η Προεδρία λοιπόν η Ιταλική θα αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της δράσης της στην καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Πρόκειται προφανώς για φαινόμενα τα οποία υποβιβάζουν, απαξιώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πολλές φορές τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις πρακτικές τις οποίες έχουμε και να διαχείσουμε καλύτερα τις βέλτιστες πρακτικές, ιδίως για να προστατεύσουμε τα παιδιά και από το φαινόμενο της εξαφάνισης. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεργαστούν από κοινού για να βρουν συγκεκριμένε απαντήσεις στις προκλήσεις αυτές, καθώς επίσης και συναδειόμενες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς αυτό, Όσον αφορά δηλαδή τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε το ακόλουθο. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, σε καμία περίπτωση στο παρελθόν δεν υπήρξε καμία τέτοια ομοσπονδία κρατών η οποία έχει καταργήσει τα εξωτερικά σύνορα με τον τρόπο που εμεί το κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Σέγγεν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε λοιπόν να έχουμε την καλύτερη εσωτερική διαχείριση των συνόρων και παράλληλα να έχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Αυτό ακριβώ κάναμε. Καταργήσαμε εσωτερικά τα σύνορα, αλλά από την άλλη από κοινού αποφασίσαμε να διαχειριστούμε συλλογικά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταβάλουμε λοιπόν εμείς περαιτέρω προσπάθειες για κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν κατά προτεραιότητα. Συγκεκριμένα λοιπόν μέτρα προκειμένου να εφαρμόσουμε τα συμπεράσματα της Task Force για τη Μεσόγειο. Θα πρέπει να καταφέρουμε να ενισχύσουμε το προσωπικό αλλά και τη χρηματοδότηση της Frontex προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στην υπηρεσία αυτή να διαδραματίζει πιο σημαντικό ρόλο στο Μεσόγειο αλλά να καταφέρουμε επίσης να δώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση στην επιχείρηση Mare Nostrum. Κάθε φορά που μιλάμε για σύνορα δεν αναφερόμαστε μόνο στις, στα μεσογειακά προφανώς σύνορα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικά είναι και τα σύνορα κάθε φορά που μιλάμε για την ανατολική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλα τα μέσα τα οποία μας παρέχει η Eurosur προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα όμως θα πρέπει να προωθήσουμε και την ανάπτυξη ενός συστήματος νόμιμης μετανάστευσης, νόμιμες οδοί μετανάστευσης δηλαδή, για τους μετανάστες εκείνους που καλή την πίστη έρχονται να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ζήτημα αυτό το αναφέραμε και στην άτυπη σύνοδο του Μιλάνου. Είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο έντονη συνεργασία ανάμεσα στην εσωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε ένα Συμβούλιο ΔΕΗ το οποίο να συνεδριάζει με το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων θα προωθήσουμε περισσότερο τις πρωτοβουλίες ελληνικής προεδρίας όσον αφορά το πακέτο για τεφή σύνορα, θα προωθήσουμε ένα νέο κώδικα για τις θεωρήσεις, καθώς επίσης και την δημιουργία ενός νέου κανονισμού για τις θεωρήσεις νόμιμης κυκλοφορίας των μεταναστών. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε περισσότερο την οδηγία για την νόμιμη εισδοχή μεταναστών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ζητήματα έρευνας και πανεπιστημιακής κατάρτισης. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε περισσότερο την αμοιβαία αναγνώριση των ανθρώπων που υπόκειται στο σύστημα διεθνούς προστασίας. Όσον αφορά τώρα το άσυλο, προφανώς πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για το άσυλο και μια κοινή στρατηγική, σφαιρική στρατηγική για το ζήτημα αυτό. Το άλλο, ο άλλος σημαντικός πυλώνος όμως πέρα από το άσυλο είναι η ίδια η ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω αυτή τη στιγμή, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι η ασφάλεια αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. αφού είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ίδιες ευρωπαϊκές μας αρχές. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε την εσωτερική στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ιταλική Προεδρία προτίθεται να κάνει εδώ πέρα μια πολύ σημαντική αναθεώρηση. Θα πρέπει να καταφέρουμε να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, παράλληλα όμως αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα εσωτερική ασφάλειας και σε σχέση με τις τρίτες χώρες θα πρέπει να καταβάλουμε πολύ σημαντικές προσπάθειες γιατί η αναθεώρηση της στρατηγικής αυτής για την εσωτερική ασφάλεια θα πρέπει να ελοποιηθεί μέσω συγκεκριμένων συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε αυτό να γίνει μέχρι τα τέλη του 2014. Η συνεργασία επίσης των αστυνομικών αρχών καθώς επίσης και της Ευρωπόλου μπορούν να συμβάλλουν πάρα πολύ στο στόχο αυτό. Όσον αφορά τώρα πάλι τις προτεραιότητές μας, ένα άλλο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι η παρίσφρηση παράνομων εγκληματικών οργανώσεων στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα μας απασχολήσει λοιπόν στην εδράση που θα έχουμε για την καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων, ιδίως όταν αυτές παρισφρίουν στις δημόσιες συμβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προωθήσουμε την καταπολέμηση της διαφθοράς και την καταπολέμηση προφανώς της τρομοκρατίας. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και θα πρέπει προφανώς να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα το φαινόμενο των μεμονωμένων τρομοκρατών, lone wolves, καθώς επίσης και το φαινόμενο των ξένων μαχητών, foreign fighters. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την καταπολέμηση ειδικών μορφών εγκληματικότητα, τα εγκλήματα βία δηλαδή, τα εγκλήματα που βασίζονται στι διακρίσει με βάση το φύλλο και την βία κατά των γυναικών. Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θα αφιερώσουμε εδώ πέρα πάλι πολύ σημαντική εργασία. Και τέλο, ξεκινώντα με το άτυπο συνέδριο του Μιλάνου, προσπαθήσαμε να θέσουμε στα πλαίσια των προτεραιοτήτων μα το ζήτημα τη προστασία των πολιτών και ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το ζήτημα της πρόληψης των καταστροφών Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές ε, αντιμετωπίζεται μονομένα από κάποιους υπουργούς ε, εξωτερικών, άλλες πάλι φορές αντιμετωπίζεται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο από συγκεκριμένε αρχές. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η συζήτηση να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για άλλη μια φορά σας λέω ότι θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια περίοδο πολύ ψηλής ευθύνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θεωρώ ότι βρισκόμαστε ήδη και σε ένα στάδιο ο επικοδομητικής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε και εμείς ως Συμβούλιο να συμβάλλουμε σε μια πιο ασφαλή και ελεύθερη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Αντζελίνο. Και ευχαριστώ και για την τήρηση του χρόνου. Ξέρω ότι είχατε πάρα πολλά να πείτε, αλλά καταφέρατε να ε, χωρέσουν στον χρόνο που είχατε. Ευχαριστώ πολύ περάσουμε αμέσως στον Υπουργό κύριο Ορλάντο για να μας παρουσιάσει τις προγραμματικές δηλώσεις και τις προτεραιότητες από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Μωράες. Να σας ευχαριστήσω επίσης για τη συμβολή σας στην άτυπη αυτή σύνοδο του Μιλάνου και να βέβαια χαιρετήσω και όλα τα μέλη της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής σας αυτής, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Θα ήθελα καταρχάς να ευχηθώ Καλή εργασία στην Επιτροπή αυτή, η οποία συστάθηκε πριν από μερικέ ε, μέρε. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πολύ ε, σημαντική νομοθετική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει από κοινού να ξαναδούμε τι ε, πολιτικέ, τι κοινοτικέ, τι οποίε θα προωθήσουμε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία αυτή, κατά τη διάρκεια τη κοινοβουλευτική αυτή θητεία. Ξεκίνησε την πορεία της και η Ιταλική Προεδρία. Θα ήθελα λοιπόν να σας διασφαλίσω, να σας επιβεβαιώσω, με συγχωρείτε όπω είπε και ο Υπουργό Ορλάντο, ότι επιθυμώ και εγώ να έχω μαζί σα την καλύτερη δυνατή συνεργασία όσον αφορά τον τομέα τη αρμοδιότητά μου, δηλαδή τα ζητήματα δικαιοσύνη. Και αυτό κατά τη διάρκεια όλου αφού του εξαμήνου τη Ιταλική Προεδρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ενισχύσουμε περισσότερο τη συνεργασία αυτή. Ο στόχο τη ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνη με, την πλήρη, με τον πλήρη σεβασμό των θεμελιώδων δικαιωμάτων και λαμβάνοντα υπόψη βέβαια και την εθνική δικαιοδοσία και νομοθεσία των κρατών μελών αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Θέλουμε να προωθήσουμε την πολιτική αυτή σε όλους τους τομείς, στο, στα πλαίσια του αστικού και του ποινικού δικαίου, στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, καθώς επίσης και στην καλύτερη δυνατή κατάρτιση των δικαστικών. Ξέρω ότι για το ζήτημα αυτό υπήρξε μια πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια του άτυπου Συμβουλίου ΔΕΗ. Θεωρούμε ότι η κατάρτιση των δικαστικών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, εφόσον μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα δικαιοσύνη και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο τι κοινοτικέ μα πολιτικέ. Η Ιταλική Προεδρία δίνει ιδιαίτερη σημασία επίση στι στρατηγικέ κατευθυντήριες γραμμέ για το χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Και εκμεταλλευόμαστε επίση ε, την ευκαιρία αυτή τη άτυπη συνόδου του Μιλάνου και θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον πρόεδρο Μωράη, προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε την άμεση εφαρμογή αυτών των ε, κατευθύνων γραμμών σε νομοθετικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον χώρο αυτό. Ως προς αυτό λοιπόν αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τρεις βασικούς τομείς, τις δικονομικές εγγύσεις, με συγκεκριμένες απαιτήσεις που απορρέουν και αποδίδεται τη συνθήκη της Λισαβόνα, προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε περισσότερο τα δικαιώματα των υπόπτων, θέλοντας να προωθήσουμε περισσότερο την προσέγγιση του Τάμπερε, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε πιο αποτελεσματικές έρευνες και δίκες. Θέλουμε επίσης όμως να προωθήσουμε περισσότερο την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και η ίδια Ιταλική Προεδρία λέει ότι θα πρέπει να επεκταθεί η αμοιβαία αυτή αναγνώριση και να αναγνωρίζουμε επίσης αμοιβαίως και τις αποφάσεις κατά σχέσεων καθώς επίσης και τις αποφάσεις κατά των εγκληματικών οργανώσεων που παρισφρίουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλουμε όμως και τις ε, την απαραίτητη συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να μπορούν και τα εθνικά δικαστήρια να γνωρίζουν καλύτερα ποια είναι τα κοινοτικά μέσα, τα πολύπλοκα βέβαια, τα οποία έχουν πολύ συχνά στη διάθεσή του. Συντοπίσαμε, όπω και πάρα πολλά κράτη-μέλη, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διασύνδεση ανάμεσα στου εξή τρίτου τομεί. Το να καταφέρουμε να έχουμε μια αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων, προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στι διαφορετικέ δικαστικέ αποφάσει που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι κανόνε προφανώ, αλλά και η εμπιστοσύνη η οποία θα πρέπει να απορρέει από τους νέους αυτούς κανονισμούς που αφορούν το δικαστικό σύστημα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Υπάρχει μια διασύνδεση προφανώς μεταξύ των κρατών μελών, αλλά η διασύνδεση αυτή θα πρέπει να μην περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένου τομείς πολιτικής, αλλά θα πρέπει να επιτυγχάνεται και στον τομέα της δικαιοσύνης. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις επόμενες ημέρες θα έχω μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Ράιχτερ η οποία πριν από λίγε μέρες ανέλαβε την αρμοδιότητά της αυτή, προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στους βασικούς στόχους του προγράμματος Ιταλικής Προεδρίας, ιδίως στους τομείς που αφορούν τη δική σας την ε, Επιτροπή και θα ήθελα επίσης να βαθύνω λίγο περισσότερο στη συνέχεια και σε ερωτήσεις που ενδεχομένως να υποβάλλετε, προκειμένου να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά τα συστήματα δικαστικής συνεργασίας, θα έχουμε μία στενή διασύνδεση ανάμεσα στις πολιτικές της δικαιοσύνης και τις πολιτικές συνερικών υποθέσεων, καθώς επίσης και μια σημαντική διασύνδεση με το ζήτημα της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Όπως είπε και ο Υπουργό Αλφάνο, θα καταπολεμήσουν οποιαδήποτε εγκληματική παρίσφρηση στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προωθήσουμε επίσης ένα διάλογο με τις τρίτες χώρες στον τομέα της δικαιοσύνης και των συνερικών υποθέσεων για κάποιους τομείς που μας ενδιαφέρουν από κοινού, για παράδειγμα καταπολέμηση εγκληματικότητας, η καταπολέμηση διακίνησης ε, ε, ανθρώπων, καθώς επίσης και τα πολέμηση της τρομοκρατίας. Θα ασχοληθούμε όμως επίσης και με το ζήτημα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και με το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της επεξεργασίας τους. Τα ζητήματα αυτά αναφέρθηκε και ο Υπουργός Αλφάν. Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο προσπάθησε να δημιουργήσει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Ιταλική λοιπόν Προεδρία καταβάλει προσπάθειε προκειμένου να υπάρχει μια συνεκτικότητα ανάμεσα στο γενικό αυτό καθεστώ και τι συγκεκριμένε παρεμβάσει που μπορούν να γίνουν στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων τη δικαιοσύνη. Προβλέπουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε την πρόοδο που ήδη έχει σημειωθεί στην ανταλλαγή των προσωπικών αυτοδεδομένων και στην επεργασία των δεδομένων αυτών τόσο σε γενικό επίπεδο όσον αφορά και στη συγκεκριμένη χρήση του στι δικαστικές διαδικασίε. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον κατάλληλο συντονισμό ανάμεσα στα δύο αυτά μέσα και θα καταφέρουμε να πετύχουμε το καλύτερο επίπεδο προστασίας καθώς επίσης και το καλύτερο επίπεδο συντονισμού ανάμεσα στις διάφορες δικαστικές αποφάσεις. Είναι πολύ σημαντικό όμω να έχουμε και μια επικοδομητική ανταλλαγή δεδομένων με τι τρίτε χώρε, ιδίω για ζητήματα επιβολή του νόμου και πρόληψη σοβαρών εγκλημάτων. Θα δώσουμε επίση ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία ενό συστήματο έντονη προστασία των προσωπικών αυτοδεδομένων δεδομένων και σε άλλα νομοθετήματα, με συγχωρείτε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται ιδιαίτερα, το γνωρίζουμε το ζήτημα αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να συμβάλλει έτσι ώστε σε πρώτη ανάγνωση να καταφέρουμε να εγκρίνουμε τη σχετική αυτή πρόταση. Συζήτησαμε ήδη με τον εισηγητή σα, τον κύριο Άλμπρεχτ, ο οποίο ήταν αντιπρόεδρο τη Επιτροπή σα, και καταφέραμε να συμφωνήσουμε στι ε, νέε αυτέ ρυθμίσει που θα πρέπει να ισχύουν για το ζήτημα τη ιδιωτική ζωή, που θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδε δικαίωμα. Θεωρούμε επίση ότι θα πρέπει να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ε, δικαστική και νομική ασφάλεια όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης θα πρέπει οι Ευρωπαίοι νομοθέτες να λάβουν υπόψη και την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ήδη έχει αποφανθεί για το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα τον ποινικό τομέα, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της σύστασης Ευρωπαϊκής Αγγελίας θεωρούμε ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ στη δημιουργία ενός γνήσιου χώρου ευρωπαϊκής δικαιοσύνης θα πρέπει να σημειώσουμε πολύ σημαντική πρόοδο στο φάκελο αυτό, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό νέο θεσμικό όργανο, το οποίο θα είναι σε θέση να διερευνά, να διώκει ποινικά και να παραδίδει ενώπιον τη δικαιοσύνη ε, του εγκληματίε εκείνου οι οποίοι ζημιώνουν ε, τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω η ευρωπαϊκή αυτή συγγελία να έχει συγκεκριμένε αρμοδιότητε, να οριοθετείται ακριβώ ο ρόλο του σε σχέση με του εθνικού δικαστέ, να γνωρίζει ακριβώ σε ποιο πλαίσιο μπορεί να λάβει δράση. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει καταφέρει να ενισχύσει και την προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ως προς αυτό στο Μιλάν ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αφαιρθούμε περισσότερο στις ερευνητικές αρμοδιότητες που θα έχει η ΕΠΟ, η Ευρωπαϊκή δηλαδή Εισαγγελική Αρχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβάλλει όμως η συζήτηση αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταφέρουμε να μειώσουμε και το χάσμα αυτή τη στιγμή απόψεων που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα όμως από τον κανονισμό ΕΠΟ Θέλουμε επίσης να υποβάλουμε στην προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την αναγκαιότητα να ξεκινήσουμε άμεσες διαπραγματεύσεις όσον αφορά το ζήτημα της ενίσχυσης των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε επίσης και τη Eurojust. Κατά αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε τη δράση της και θα της επιτρέψουμε να ενισχύσει την εργασία της Ευρωπαϊκής Αγγελία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να, να διασυνδέσουμε περισσότερο τα τρία αυτά ζητήματα. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Χώρου δικαιοσύνης και εφαρμογή της, του κανονισμού εκείνου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε λοιπόν μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία θα μπορεί να κάνει τις απαραίτητες έρευνες και να καταπολεμά κατά αυτόν τον τρόπο την απάτη εναντίον του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποτελεί μια πραγματική προστιθέμενη αξία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε οποιαδήποτε επικάλυψη. Όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων στα πλαίσια των ποινικών υποθέσεων, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για τι δικονομικέ εγγυήσει για του ανήλικου. Ήδη ξεκινήσαμε μία σχετική εξέταση στο Συμβούλιο όσον αφορά το τεκμήριο αθωότητα και το ευεργέτημα παινία. Μόλις η Επιτροπή σας διορίσει εισηγητή για τα ζητήματα αυτά θα μας σε θέση να ξεκινήσουμε επικοδομητική συνεργασία μαζί σας. Η καταπολέμηση τώρα των διαφόρων μορφών εγκληματικότητας, η εμπορία δηλαδή των ανθρώπων, καθώς επίσης και η διεθνής διεθνική εγκληματική δράση αποτελεί ζήτημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη και προφανώ την Προεδρία μα. Και πειράζει προφανώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καθώ επίση και την κοινωνία των πολιτών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια έντονη πολιτική διάσταση στην πρόκληση αυτή. Οι εγκληματίε και οι εγκληματικέ οργανώσει θα πρέπει να μην έχουν πρόσβαση σε κανένα έσοδο από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα. Ω προ αυτό λοιπόν, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ε, πρόθεσης, της συζήτησης της ε, αρχής ε, της αμοιβαία αναγνώρισης, η οποία θα πρέπει επίσης να ισχύει και για τις διάφορες δικαστικές αποφάσεις όσον αφορά οποιαδήποτε μορφή κατάσχεσης και δίμευσης των εγκληματικών προσόδων. Μάλιστα το ζήτημα αυτό θα μα απασχολήσει και σε σύνοδο που θα διεξαχθεί στη Σιρακούσια στι 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Και προφανώ θα θέλαμε να έχουμε και τη συμβολή τη δική σα τη κοινοβουλευτική επιτροπή. Η δημιουργία μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή αποτελεί τμήμα μια στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει μέσα όλο και πιο πολύπλοκα για τη δικαστική συνεργασία στον τομέα των ποινικών και στον τομέα των αστικών. Και θέλουμε λοιπόν να έχουμε και την κατάλληλη κατάρτιση των δικαστικών, των δικαστών, καθώ επίση και των εισαγγελέων. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Κατάρτισης. Τέλος, θα έχουμε τις ε, συνήθεις υπουργικέ ε, διασκέψεις Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δυτικά Βαλκάνια και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε με την κυβέρνησή μας και το Υπουργείο Εξωτερικών μας μια ενδεχόμενη επανεκκίνηση του διαλόγου με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εν κατακλείδη θα ήθελα να διασφαλίσω ότι ε, η Ιταλική Προεδρία θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλε αυτέ τι προκλήσει οποίε ανέφερα προκειμένου να έχουμε ένα γνήσιο δικαστικό χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου στα πλαίσια του χώρου αυτού να μπορούν να τηρούνται απόλυτα τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών και να μπορούμε όμως να πατάξουμε τη διαφθορά, την απάτη και το οργανωμένο έγκλημα. Θέλουμε να έχουμε μια επικοδομητική, ειλικρινή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη είδαμε ότι έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε μία συμφωνία, στο προηγούμενο δηλαδή άτυπο συνέδριο, όσον αφορά την εξακρίβωση της ηλικίας των νέων μεταναστών. Πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε επίσης να προωθήσουμε περισσότερο τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και μειώνουμε επίσης κατά αυτόν τον τρόπο και την γραφειοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όχι μόνο να έχουμε μια θετική συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων, αλλά και μια πιο ειλικρινή ε, επικοδομητική συνεργασία και επαφή με τους ίδιους Ευρωπαίους πολίτες. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε τους πολίτες εκείνους οι οποίοι καλούνται να έρθουν σε επαφή με διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για το ζήτημα λοιπόν αυτών της επαφής με τους Ευρωπαίους πολίτες είμαι σίγουρο ότι η δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα συμβάλλει πάρα πολύ στο έργο το οποίο ήδη επιτελεί αυτή τη στιγμή η Ιταλική Προεδρία. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. <clears throat> Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα. Θα ήθελα να πω στα μέλη ότι ε, δεν μιλάτε μόνο εδώ για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Επανειλημμένα και στο άτυπο Συμβούλιο ε, θυμίζατε στο Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό νομοθετικό σου και πολιτικό ρόλο να διαδραματίσει και ιδιαίτερα στην προστασία των δεδομένων. Το ίδιο μήνυμα δώσατε και εδώ, αλλά το εκπέμπεται και προς το Συμβούλιο. Και καλό είναι να το γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής μας και χάρηκα πάρα πολύ που τα ξανά άκουσα. Και για την Task Force. Ε, πραγματικά είναι στην πρώτη γραμμή η Ιταλία είναι πολύ σημαντικό και αυτό το μήνυμα να περάσει. Έχουμε πολλά έμπειρα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Πολύ μακρύς κατάλογο κατάλογος των ομιλητών. Παρακαλώ, θέλω να δώσω το παράδειγμα να μην μιλήσω πολύ ώρα. λέω στα νέα μέλη ότι για να ζητούν το λόγο πρέπει να σηκώνουν το χέρι τους ή το καρτελάκι με το όνομά τους για να σημειώνει η γραμματεία ότι θέλετε το λόγο για να σας δοθεί στη συνέχεια αφού εγγραφείτε στον κατάλογο. Πρώτοι όμως οι ε, συντονιστές. Είναι πάρα πολύ μακρύς ο κατάλογος όπως μπορείτε να φανταστείτε. Παρακαλώ λοιπόν όλοι να περιοριστείτε όσο μπορείτε. Και επίσης να μας λέτε και σε ποιον υπουργό απευθύνετε την ερώτησή σας για να μπορέσουν να μοιραστούν ε, τις απαντήσεις και παρακαλώ να κάνετε ερωτήσεις και όχι σχόλια ή τοποθετήσεις. Πρώτη η κυρία Χολμάιερ και μετά ε, κυρία Σίπελ. Η Μόνικα πρώτη Χολμάιερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πραγματικά θα περιοριστώ σε ερωτήσεις, δεν θα κάνω ούτε σχόλια, ούτε παρατηρήσεις, ούτε ε, τοποθετήσεις και ιστορίες. Θα τα ξαναπούμε αργότερα αυτά στην Επιτροπή, έχουμε όλη την ευχαίρεια. Θα ήθελα καταρχάς να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό, τον κύριο Αλφάνο. Η Ιταλία, όπως και άλλες χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, αντιμετωπίζει τεράστιο κύμα μετανάστευσης, όπως ε, ακούω και από τα κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αυξάνεται και εκεί η πίεση. Δεν περιορίζεται μόνο στη Μεσόγειο δηλαδή η κατάσταση αυτή. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μπορεί να συνεισφέρει η Ιταλική Προεδρία έτσι ώστε το θέμα αυτό να μην το αντιμετωπίζουμε μόνο ε, από τη σκοπιά, τη βραχυπρόθεσμη και των ε, οξέων προβλημάτων που έχουμε τώρα για να προτείνουμε καταστάσεις και λύσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά να έχουμε μια ευρεία εποπτεία στη συνεργασία με την εξωτερική πολιτική, πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας, μέτρα εσωτερικής πολιτικής και ανθρωπιστική βοήθεια, για παράδειγμα. Δηλαδή, ε, να διαρθρώσουμε και να συνδέσουμε την όλη μας συνύπαρξη και συλλειτουργία με αυτά τα μέρη του κόσμου. Η Ιταλική Προεδρία μπορεί να θέσει ένα κάποιο πλαίσιο και να βοηθήσει στην εκπόνησή του μαζί με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συζήτηση. Και ένα δεύτερο που αναφέρατε ήταν η συνεργασία και σε επίπεδο Frontex και ε, ανάπτυξη και διεύρυνση του οργανισμού. Ποιες είναι οι επιθυμίες και τα μέτρα που θεωρείτε εσείς σκόπιμα για το Frontex ε, και απαραίτητα και να κάνουν τα διάφορα κράτη ανεξαρτήτως γεωγραφικής τους θέσης για να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Ένα δεύτερο που αναφέρατε ήταν η τρομοκρατία. Ε, τι είδους πρωτοβουλίες προβλέπει η Ιταλική ε, Προεδρία και προγραμματίζει σχετικά με αυτό. Γιατί έχουμε και την κατάσταση του ε, ίσης και τους λεγόμενους ξένους μαχητές που επαναπατρίζονται και είναι ε, καινοφενή αυτά τα ζητήματα. Ε, ο ίσως είναι ο Ισραμικό στρατός στο Ιράκ και στη Συρία. Ε, το Ισραμικό κράτος, συγγνώμη. Και για την κατανομή των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχω λίγο την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ στοιχειώδεις οι αρμοδιότητες αυτές ενώ όταν πρόκειται για πολύ βαριά εγκληματικότητα διασυνοριακού χαρακτήρα σχεδόν δεν έχει καθόλου ουσιαστικέ αρμοδιότητες. Επιπλέον έρχομαι να διαπιστώσω ότι στη Eurojust δεν υπάρχει αύξηση της ε, χρηματοδότησης. Οπότε εκεί πώς φαντάζεστε την ε, εργασία ενός Ευρωπαίου εισαγγελέα και οικονομικά αλλά και γενικότερα με ουδετερότητα ως προς τον προπολογισμό, δηλαδή όχι αύξηση των κονδυλίων. Είναι κάπως δυσχερής αυτή η λειτουργία. Θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε αυτό και ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει μια πρόσφατη απόφαση του ΔΕΚ για την προληπτική ε, διατήρηση ε, και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων. Η Ιταλική Προεδρία τι ε, προτίθεται να ε, αναλάβει ως πρωτοβουλίες για να υπάρχει κάποια στοιχειώδης συνάφεια και συνέχεια στις πολιτικές των κρατών μέλων. Ευχαριστώ Μόνικα. Παρακαλώ για τελευταία φορά. Μάλλον ε, τώρα που είπα να ζητήσετε το λόγο, ζήτησαν το λόγο όλα τα μέλη της Επιτροπής. Μήπως δεν θα πρέπει να σας αθαρρύνω τόσο πολύ και να είμαι λίγο πιο δικτυοποιητικός Γιατί έχει τριπλασιαστεί πλέον ο κατάλογος σε μέγεθος. Ε, παρακαλώ για να μην έχουμε απογοητευμένους ε, ε, βουλευτές και να ε, μπορέσει να ξανάρθουν και οι υπουργοί <laughs> κάποια στιγμή για να απαντήσουν. Λοιπόν, οι συντονιστές επαναλαμβάνω και οι υπόλοιποι όσο γίνεται πιο σύντομα. Αλλά να είστε όσο γίνεται συντονιστές και τα υπόλοιπα μέλη. Ε, Μπίρκετ, είσαι επόμενη. Ε, και είσαι συντονίστε Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζίπελ. Θα ήθελα και εγώ να αρχίσω με ερωτήσεις. Έχω μερικές ερωτήσεις προς τον Υπουργό κύριο Αλφάνο. Πρόκειται πάντα για την πολιτική μετανάστευσης και εγώ διερωτώ με. Συγκεκριμένα, πώς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που είναι υποχρεωμένοι να φεύγουν από τον τόπο τους, έχουμε πρόσφυγες από τη Συρία, Φερρυπίν, αυτοί ουσιαστικά πώς θα μπορέσουν να, μπορούν να φτάνουν στην Ευρώπη και να κάνουν αίτηση ασύλου, να είναι δεδομένη αυτή η δυνατότητα εφόσον από την άλλη πλευρά μιλάμε όλο και περισσότερο για την ασφάλεια των συνόρων, για τη φύλαξη. Βεβαίως θα πρέπει να φύλουμε τα σύνορά μας, αλλά όλο μιλάμε για αύξηση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Frontex. Πολύ συγκεκριμένα εσείς πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι άνθρωποι που είναι πρόσφυγες και έχουν ανάγκη να μπορούν να βρουν ένα λιμάνι καταφυγής και να κάνουν αίτηση ασύλου ακόμα και αν είναι υποχρεωμένοι για να φτάσουν σε αυτό το λιμάνι να καταφύγουν στις υπηρεσίες ενός δουλεμπόρου γιατί δεν ξέρουν πώς να φύγουν από τη χώρα τους για να πάνε σε άλλη χώρα και απευθύνονται σε αυτούς τους διακινητές. Και επίσης ένα άλλο ερώτημα. Η πίεση στα σύνορα, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, είναι αφόρητη και για να χαλαρώσει αυτή τίθεται το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης, γιατί όλοι οι πρόσφυγες δεν είναι πρόσφυγες με την κλασική έννοια της χορήγησης ασύλου, είναι και μετανάστες. Ε, θέλουμε και μπορούμε με τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να ανοίξουμε αυτή τη δυνατότητα για να επιτραπεί η νόμιμη μετανάστευση και πώς αυτή θα οργανωθεί. Θα υπάρξουν, ε, ξέρω κι εγώ, ε, ποσοστώσεις, θηρίδες που πρέπει να απευθύνουν γίνεται κάποιος μέχρι τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται μικρά βήματα για την εποχιακή εργασία, ε, μια αντίστοιχη οδηγία ή άλλα μικρομέτρα, μεσοβέζικες λύσεις, δεν είναι λύση αυτό για ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση. Έχω και δύο ερωτήσεις όμως προς τον Υπουργό κύριο Ορλάντο. Αρχίζω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις εδώ. Εάν θα πρέπει να είναι αρμόδια για πάρα πολλά κακουργήματα ή εγκλήματα ή μόνο για ε, αξιόπινες πράξεις που προσβάλλουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου πολιτική ομάδα και εγώ προσωπικά ήμασταν υπέρ αυτού του περιορισμού, γιατί δεν μπορούσαμε να φανταστούμε καθόλου σε ποιο νομικό πλαίσιο μπορεί να δουλέψει μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ιδιαίτερα ε, όταν αυτό αφορά περισσότερα από ένα κράτη-μέλη. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που ισχύει, ε, ποια είναι η δικαιοδοσία, σε ποιο δικαστήριο θα πάνε, ε, τι δικαιώματα έχουν οι κατηγορούμενοι, ποιε είναι οι κυρώσει που επιβάλλονται, όλα αυτά πώ θα ρυθμίζονται. Γι' αυτό στην αρχή εμείς θεωρούσαμε ότι θα πρέπει σε πρώτη φάση να περιοριστεί η δουλειά ε, του εισαγγελέα να δοκιμαστεί πριν δημιουργήσουμε τελεσμένα γεγονότα που ε, είναι πανάκριβα και καθόλου αποτελεσματικά. Και ένα άλλο ακόμα εδώ για την προστασία δεδομένων. Γιατί στο θέμα του ε, Ευρωπαίου εισαγγελέα τίθεται το θέμα της συνεργασίας αστυνομικών και διοκτικών και δικαστικών αρχών και υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις για τις αστυνομικές έρευνες, για τη συλλογή ε, αποδεικτικών στοιχείων, πιστήριων, πώς αυτά τηρούνται, πώς αυτά την χάνουν χειρισμών. Υπάρχουν θεμελιώδη δικαιώματα και των κατηγορουμένων και των μαρτύρων και των θυμάτων και θα πρέπει να τηρούνται αυτά παντού και να γίνονται σεβαστά. Και κάτι ε, ως προς τα δικονομικά δικαιώματα ανεξαρτήτως ε, Ευρωπαίου Αγγελέα. Ε, η Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν έχουμε μόνο ως μέλημα τη βελτίωση της προστασίας αλλά και για καλά δικαιώματα και εγγυημένα δικαιώματα. Γιατί γι' αυτά δεν έχουμε λεφτά, μόνο για την προστασία. Και χρονικά πώς το βλέπετε, θα τολμήσετε να αναφέρετε η ημερομηνία για το πακέτο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα προλάβετε μέσα στο χρόνο. Ευχαριστώ, Μπρικίτ. ο συντονιστής ε, της ε, ομάδας του ECR, ο οποίος θα μας αποδείξει πόσο σύντομα μπορεί να μιλούν οι Άγγλοι, ελπίζω. Νομίζω ότι θα δείξω ότι τι μπορεί να προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι η Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μιλήσω και λίγο για θέματα ασφάλειας δεδομένου ότι πιστεύω ότι ε, η πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, ανησυχούν συνολικά για την ασφάλεια που έχουν ή δεν έχουν σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο. Στις ερωτήσεις μου θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν ε, συνεχίζω από μια προηγούμενη ερώτηση. Εξαιρετικά ασταθής είναι η κατάσταση που επικρατεί σε πολλά μέρη με τα οποία συνδέεται η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή κυρίως στη Μέση Ανατολή η αυξανόμενη δύναμη ομάδων όπως η ISIS ε, θα πρέπει να μας ανησυχεί, ή μας ανησυχεί και θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Προεδρίας για την αύξηση ή τη βελτίωση ε, στον τομέα ανταλλαγής δεδομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ποιο βαθμό θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτό στη διάρκεια της Προεδρίας, όπως επίσης και στο θέμα των Ευρωπαίων ξένων μαχητών που αναφέρθηκε έχετε καλές και ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά με αυτό. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ένταρμα Σύλληψης, η μεταρρύθμιση και το, η επαναφορά του μου φαίνεται σημαντική προτεραιότητα. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να, δοθεί, να γίνει μια δοκιμασία αναλογικότητας και στις δύο πλευρές και επίσης περισσότερες ε, διασφαλίσεις έτσι ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης σε ένα για μένα χρήσιμο εργαλείο. Το δικαίωμα τώρα στην ε, λύθη. Ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχουν ε, έρθει στην προσοχή μας πολλά παραδείγματα μεταξύ των οποίων πολλοί πολιτικοί, πολιτικών που θέλουν να αφαιρεθούν ε, αναφορές στην πολιτική τους, ε, που τους κάνουν επικρίσεις ή εγκληματίες που ζητούν άρθρα και επίσης ε, διάφοροι που έχουν μετανιώσει για αυτό που έχουν ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βεβαίως η κρίση, η δικαστική κρίση είναι κατά τη γνώμη μου διατυπωμένη με ασαφή τρόπο και πρέπει να φροντίσετε να κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε η δικαστική απόφαση που έχει σχετικά ληφθεί να μην ε, περιορίσει την προστασία της ασφαλείας μας. Ασυνόδευτη ανήλικη. Θα ήθελα να ακούσω την Επιτροπή, την Επιτροπή που να μας πει τι έχει σχέση, τι σκοπό να κάνει σε σχέση με την εξαιρετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε στην περασμένη θητεία. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το θέμα, ανησυχώ πολύ για την ταχύτατη αύξηση του αριθμού ανθρώπων πολύ μικρών παιδιών που ή χρησιμοποιούνται ή κακοποιούνται και που σαφώς αντιμετωπίζονται από ανθρώπους που δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη τους. Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί πραγματικά έσχος για θα πρέπει να, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί ταχύτατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Συντονιστής της, συντονίστρια της ομάδας Άλντε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο υπουργούς που ήρθαν σήμερα εδώ. Να αναφερθώ στο θέμα της μετανάστευσης που αναφερθήκατε, στο οποίο αναφερθήκατε εσείς κύριε Αρφάνου. Βεβαίως όλα αυτά με βάση την ε, τραγωδία στην Λαμπετούσα το περασμένο Οκτώβριο που χάθηκαν πάνω από 360 ζωές. Αλλά τέτοιες τραγωδίες συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά, κάθε εβδομάδα και οι πολίτες της Ιταλίας διασώζουν τους ανθρώπους αυτούς. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να τους ευχαριστήσω, να αναγνωρίσω αυτό το οποίο κάνουν. Κύριοι Υπουργοί, αναφερθήκατε στα θέματα της Frontex, της επιβολής του νόμου, στον έλεγχο των συνόρων κλπ. Αλλά κάτι στην ε, έλειπε πάρα πολύ από την ομιλία σας το γεγονός ότι κάθε σημερινός ε, μετανάστης είναι παράτυπος δεδομένου ότι δεν υπάρχει ασφαλής ε, νόμος τρόπος ένταξης στην Ευρω... Ε, εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε λοιπόν να σας ρωτήσω, τι σκοπεύετε να κάνετε αν κάτι, οτιδήποτε στη διάρκεια της Προεδρίας σας, τι σκοπεύετε να φέρετε στην επιφάνεια ώστε να υπάρξουν νόμιμοι και ασφαλή δρόμοι για αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από την διώξη και να, που έχουν δικαίωμα σε διεθνή προστασία στην Ευρώπη, στις χώρες μας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενέβης. Τι σκοπεύετε να κάνετε και αν δεν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, παρακαλώ να μας το πείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σίλια συντονιστής της, ομάδα, της συντρόφισης ομάδας Η κυρία Κορνέλη Ευχαριστώ. Τρεις ενότητες ε, ερωτήσεων. Η πρώτη απευθύνεται και προς τους δύο υπουργούς. Τώρα πέντε χρόνια είχαμε το λεγόμενο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για τα εσωτερικά και τη δικαιοσύνη. Μια ε, πενταετία μας απασχόλησε, διάφορα μέτρα και πρωτοβουλίες ελήφθησαν. Ερωτώ λοιπόν και τους δύο υπουργούς. Θα αγωνιστείτε ε, για μια λογική αξιολόγηση και ένα απολογισμό αυτού του προγράμματος ή θα προτείνετε συνεχώς νέα προγράμματα που έρχονται να προσθεθούν. Ε, θα γίνει καμία αξιολόγηση του όλου εγχειρήματο ή όχι. Το δεύτερο, προστασία δεδομένων. Ερωτώ τον Υπουργό Ορλάντο. Με έχει ενοχλήσει λίγο αυτό που είπατε. Μιλήσατε για ε, μέγιστη προστασία δεδομένων αφενός, αφετέρου, λέτε ότι είναι, ε, θα πρέπει να είναι όσο γίνεται αποτελεσματική αυτή, επανειλημμένα. Για το πακέτο αυτό καθ' αυτό δεν είπατε σχεδόν λέξη, ε, για να μπορέσουμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Αρχίζω από την οδηγία, που είναι το αποπέδι του Συμβουλίου. Ε, πώς έχει αυτή η κατάσταση σήμερα. Μιλώ για ένα θέμα που αφορά την Ευρωπόλ και άλλα ποια είναι η διάθεση του Συμβουλίου. Ε, ασχολείται με αυτό, δουλεύει. Το δεύτερο για την προστασία των δεδομένων αφορά βεβαίως τον κανονισμό. Θα ήθελα να πω ότι στην προστασία δεδομένων το θέμα δεν είναι μόνο να εξασφαλίζουμε ε, την προστασία των δεδομένων ή την ανταλλαγή τους για θέματα εγκληματικότητας, πρόκειται και για ιδιώτες, των οποίων τα στοιχεία ε, ανταλλάσσονται και θα πρέπει να προστατεύονται. Λοιπόν, ρωτώ, πώς το βλέπετε αυτό. Τι θα γίνει τους επόμενους μήνες για τον κανονισμό. Πώς έχουν τα πράγματα ε, στα επιμέρους θέματα. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είπατε ότι σας ενδιαφέρει πολύ να υπάρξει συνεργασία με τρίτες χώρες. Να συμπληρωθεί, να βελτιωθεί και συγκεκριμένα τι εννοείτε. Γιατί όταν ακούω για τρίτες χώρες μου ανάβουν διάφορα λαμπάκια γιατί έχουμε τεράστια προβλήματα εκεί. Και τι, ε, μιλάτε, μιλάτε για την προληπτική διατήρηση. Θα κάνετε εκεί δηλαδή ε, προτάσεις, πρωτοβουλίες για να συλλέγονται και να διατηρούνται για προληπτικούς σκοπούς. Και κάτι άλλο για τους μεθοριακούς ελέγχους και τη μετανάστευση. Πολλή λόγος έγινε για λαθρομετανάστευση, ε, ε, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση ανθρώπων. Πολλά έχουν γραφτεί και λεχτεί. Εσείς θα κάνετε τίποτα για να ενισχύσετε τα θεμελιώδη δικαιώματα όπου υπάρχουν αυτά ή να τα θεσπίσετε τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσφύγων και αυτών που ζητούν άσυλο. Ακούσαμε ένα σωρό πράγματα. Eurosur και διάφορα τέτοια ωραία που θα φτιάξετε, Frontex θα τη διευρύνετε, τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζητούν άσυλο, πώς θα εξασφαλιστούν. Ο κύριος Γιούγκερ ζήτησε εναρμόνιση του δικαίου ασύλου. Θα γίνει τίποτα κατά τη διάρκεια του δικού σας εξαμήνου προωθείτε τίποτα, υπάρχουν ε, πρωτοβουλίες και ένα τελευταίο βεβαίως σαφές. Χτες και προχτές είχαμε πάλι πνιγμούς στη Μεσόγειο. Τι θα κάνετε έτσι ώστε οι πρόσφυγες να μην χάνουν τη ζωή τους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας ε, προβληματίζει και μας συγκλονίζει όλους, όχι μόνο την τελευταία πενταετία, καθημερινά. Έχετε εκεί κάποιες προθέσεις, κάποιες πρωτοβουλίες να προωθήσετε. Ευχαριστώ. Η Σκά Κέλλερ, εξορόμαστε Πρασίνο για γιατί λείπει ο συντονιστή του. Like Απευθύνομαι στον κύριο Αλφάνο και αφορά και αυτή την ερώ... η ερώτηση τη μετανάστευση. Το πρόγραμμα που στείλατε Θέλετε να ενθαρρύνετε και να διευρύνετε τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον χώρο της μετανάστευσης. Ποιες χώρες ε, συγκεκριμένα έχετε κατά νου και κατόπιν. Να συνεχίσω σε αυτά που είπαν οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλιστές και γκοε. Η νόμιμη πρόσβαση, ούτε κουβέντα γι' αυτό στο πρόγραμμά της. Είναι σκάνδαλο, είναι φοβερό. Οι μετανάστες οι πρόσφυγες μάλλον θα πρέπει να ε, εμπιστευτούν τις ζωές τους σε ελαφρεμπόρους, σε ελαφροδιακινητές. Μιλάμε για ανθρώπους από τη Συρία που είναι προφανώς ε, πρόσφυγες και δεν έχει νόημα να τις αντιμετωπίζει η Frontex. Τι θα κάνετε λοιπόν για το θέμα της νόμιμης και ασφαλούς πρόσβασης των προσφύγων. Ως Συμβούλιο, πώς έχετε σκοπό να πιέσετε τους συναδέλφους τα άλλα κρατημέλη να έχουν θέσεις εγκατάστασης για τους πρόσφυγες. Θα κάνετε μια συνάντηση, μια διάσκεψη που θα προσφερθούν θέσεις για τους πρόσφυγες από τη Συρία. Βλέπετε ότι πολλές πολιτικές ομάδες θέλουν να ακούσουν κάτι περισσότερο από αυτού και θέλω να ε, αναγνωρίσω τις προσπάθειες που έχει κάνει η Ιταλία στο Mare Nostrum και βεβαίως αυτό το κοινοβούλιο πάντοτε ζητούσε μεγαλύτερη ελληνική εκ μέρους των κρατών μελών στο θέμα της μετανάστευσης αλλά αυτό δεν ε, αφαιρεί την ευθύνη μας να αντιμετωπίσουμε ε, τους μετανάστες και πρόσφυγες και επίσης να έχουμε ένα σύστημα ασύλου που να προσφέρει νόμιμη πρόσβαση. Ένα μεγάλο θέμα είναι το θέμα της επανεγκατάστασης Λόρα Φεράλα από την ομάδα, συντονίστρια της ομάδας EFD. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τον Υπουργό Ορλάντο. Πριν από μερικές ε, μέρες είχαμε την επέτειο της ε, σφαγής στη Δία Νταμέλιο. Προέρχομαι από την Καλαβρία, γνωρίζω ακριβώς πώς λειτουργεί η μαφία Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η μαφία επισέρχεται όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα, όχι σε συγκεκριμένε μόνο περιοχέ, συγκεκριμένε χώρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μαφιόσκε οργανώσει όλο και μεγαλώνουν, όλο και αποκτούν πιο διεθνή χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλέ φορέ ε, παρισφρίουν ακόμα και στον πολιτικό τομέα, στον τομέα τον ανώτατο διοικητικό τομέα και το καθεξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε στα πλαίσια της Ιταλικής Προεδρίας ποιες είναι οι πρωτοβολίες που μπορούν να προωθηθούν. Αναφερθήκατε εσείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει όμως κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της μαφίας, συγκεκριμένα της μαφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είχε εγκρίνει στο τέλος της θητείας του ένα συγκεκριμένο κείμενο, μια συγκεκριμένη έκθεση για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όμως τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το ποινικό δίκαιο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της μαφίας. Πώς μπορούμε πραγματικά να κατασχέσουμε και να δημεύουμε την περιουσία, τα περιουσιακά στοιχεία των οργανώσεων αυτών και πώς μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο τη διερεύνηση και την ποινική δίωξη των οργανώσεων αυτών συστήματα τα οποία ισχύουν στο Ιταλικό δίκαιο αλλά όχι στο Ευρωπαϊκό δίκαιο. Όσον αφορά τη μετανάστευση, απευθύνομαι πάλι στον Υπουργό Αλφάνο. Αναφερθήκατε στο Mare και είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία ή ακόμα και απορρόφηση του Mare Nostrum από τη Frontex. Δεν ξέρω όμως αν η Frontex έχει την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα να απορροφήσει πραγματικά το Mare Nostrum. Δεν νομίζω καν ότι έχει το απαραίτητο προσωπικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε πώς μπορεί να γίνει η ενσωμάτωση αυτή του Mare Nostrum στο Frontex. Ξέρετε ότι θα μπορούσε ακόμα και ο οργανισμός των ΗΕ να επιχειρήσει στη Μεσόγειο προκειμένου να επιλύσει κάποια από τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι εργαζόμενοι της Frontex οι οποίοι ε, ε, διακινδυνεύουν ακόμα και τη ζωή τους πολλές φορές για να διασώσουν πολίτες. Πριν από μερικές ε, μέρες είδαμε ότι πάνω από 100 μετανάστες, παράνομοι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μια βάρκα η οποία βρισκόταν στα νυχτά της Λαπεντούζα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μια πραγματική διεθνή ανθρωπιστική κρίση στην Μεσόγειο. Δεν υπάρχουν άμεσες γρήγορες λύσεις που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διεθνή κοινότητα. Η Ιταλία, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, έχει σύνορα τα οποία δέχονται πολύ έντονες μεταναστευτικές πιέσεις. Πώς μπορεί πραγματικά η Ιταλία να πετύχει μια καλύτερη συνεργασία, συντονισμό αλλά και αλληλεγγύη όσον αφορά τα νότια αυτά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να έχουμε την καλύτερη συνδρομή των χωρών της Βόρειας Ευρώπης προς τις οποίες πηγαίνουν οι περισσότεροι μετανάστες. Επίσης, όσον αφορά την παραγωγή των όπλων, πρέπει να γνωρίζουμε επίσης τι ακριβώς γίνεται με το ζήτημα αυτό, γιατί πολλές φορές το αντίτιμο στις ανθρώπινες ζωές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ τελειώνει ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων. Αυτά είναι τα καλά νέα, τα το κακά είναι ότι ακολουθούν 23 ακόμα μιλήτες. Λοιπόν, με αυτή την προειδοποίηση θα παρακαλούσα τους δύο υπουργούς να απαντήσουν. Ε, σχετικά σύντομα, μην επεκταθείτε παρακαλώ. Με την Υπουργό Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης. Η κυρία Χολμάριέρα έχει απόλυτα δίκιο όταν λέει ότι δεν έχουμε μόνο τα σύνορα της Μεσογείου, αλλά έχουμε και όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα τα οποία πλήττονται από τη μετανάστευση και ιδίω τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο τόνισα και στην παρέμβασή μου. Γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της επιτήρησης των σύνορων έχει να κάνει με το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πραγματικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια επίγουσα έκτακτη κατάσταση στη Μεσόγειο, σε όλη τη Μεσόγειο και ιδίω στην κεντρική Μεσόγειο. Θα μπορούσε όμως να προκύψει μια άλλη έκτακτη ανάγκη σε κάποια άλλα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωση, όπως έχει γίνει αλλεπάλληλα στο παρελθόν, όταν ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση έπρεπε να αντιμετωπίσουν την άφηξη μεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη από τα ανατολικά με συγχωρείτε της Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειαζόμαστε μία άμεση στρατηγική η οποία να είναι τόσο βραχυπρόθεσμη όσο και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Χρειαζόμαστε λοιπόν δράση στην Αφρική, δράση στα σύνορά μας και δράση στην ίδια την εδαφική επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως Προεδρία το μόνο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ακολουθήσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Σε αυτά πρέπει να βασιστούμε. Αυτή είναι η στρατηγική στα πλαίσια της οποίας κινούμεθα. Και βλέπουμε στα πλαίσια των συμπερασμάτων αυτών αυτόν ότι διασυνδέεται σωστά το ζήτημα της μετανάστευσης με το ζήτημα του ασύλου και της επιτήρησης των συνόρων. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε προφανώς την παράνομη μετανάστευση και να διαχειριστούμε την νόμιμη μετανάστευση και να βασιστούμε επίσης όλες αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει για να δούμε πώς μπορούμε να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ελκυστική το ζήτημα λοιπόν τη μετανάστευση του ασύλου και τη επιτήρηση των συνόρων είναι τρία ζητήματα που από κοινού συντονισμένα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της ισότιμη ανάθεσης αρμοδιοτήτων και ευθυνών στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Το λέει αυτό το άρθρο 80 τη συνθήκη, όχι η Ιταλική Προεδρία. Βάσει αυτών των αρχών πρέπει εμεί να κινηθούμε. Βάσει αυτών των αρχών πρέπει να λάβουμε δράση. Προκειμένου όμω να γίνει κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε μία διεθνή προστασία. Δηλαδή, στα πλαίσια της διεθνούς προστασίας πρέπει να αναλάβουμε μια σφαιρική πολιτική δράση ως Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κοινοτική ευρωπαϊκή λοιπόν δράση για το ζήτημα του ασύλου. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί μια δράση στα πλαίσια της οποίας θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε τόσο ευθύνες και όσο και λεγγύη. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου αποτελεί σημαντικότατη προτεραιότητα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο. Αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Προφανώ θα πρέπει να έχουμε συγκλίνουσε πρακτικέ ανάμεσα στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέει αυτό το ίδιο το Συμβούλιο και το παραλαμβάνω και εγώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οποιοδήποτε έχει το καθεστώς του πρόσφυγα να μπορεί να αντιμετωπίζει ανάλογες διαδικασίες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ευθυγράμμιση λοιπόν των καθεστώτων ουσιαστικά θα ενισχύσει και τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω επίση ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολύ σημαντική δράση πρόληψη του φαινομένου τη παράνομη μετανάστευση στην Αφρική συγκεκριμένα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση και να ενισχύσουμε μέσω συνεργασία την νόμιμη μετανάστευση. Όχι μόνο με τι χώρε διέλευση, αλλά κυρίω με τι χώρε καταγωγή. Για παράδειγμα, σήμερα η Λιβύη βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ μεγάλη αστάθεια. Είναι πολύ δύσκολο εμεί να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε τη Λιβύη. Η Λιβύη όμως αυτή τη στιγμή δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που φτάνουν από άλλες περιοχές Αφρικής. Ακριβώς με αυτές τις χώρες προέλευσης, καταγωγής μάλλον, θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τη συνεργασία μας και όχι απλά και μόνο με τη Λιβύη. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ Υπουργών Εσωτερικών και Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο και την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ακριβώς έχει αποσαφινιστεί αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο. Δηλαδή να προωθήσουμε την πολιτική more for more. Να δώσουμε δηλαδή περισσότερα δικαιώματα και να κάνουμε περισσότερες παραχωρήσεις προς τις χώρες εκείνες οι οποίες συνεργάζονται, προτίθενται να συνεργαστούν περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, χρειαζόμαστε και προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στις χώρες προέλευσης και καταγωγής των μεταναστών. Πρέπει να καταφέρουμε να ενισχύσουμε μια πιο στενή συνεργασία με, τον, με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών και ελπίζω επίσης ότι θα πρέπει να δώσουμε μια υψηλότερη χρηματοδότηση, καθώς επίση να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για το ζήτημα της ε, επιστροφής, επανεισδοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακριβώς αυτό θα αντιμετωπίσει κάπως και το ζήτημα, το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με τους μετανάστες από τη Συρία. Και αυτή τη στιγμή αναφέρομαι και σε ερώτημα μιας άλλης Ευρωβουλευτή όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία. Η αστυνομική συνεργασία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων. Ξέρετε ότι η απάντηση στις περισσότερες ερωτήσεις σας έχει να κάνει με τον καλύτερο συντονισμό και τη διαφάνεια στην πολιτική που ακολουθούν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη μέχρι στιγμής μονομένα έχουν αναλάβει κάποιες αποφάσεις, δεν έχουν τις ίδιες ανησυχίες, δεν έχουν την ίδια ευαισθησία, επομένως πολλές φορές δεν συγκλίνουν τα μέτρα τους αυτά, δεν συγκλίνει η πολιτική τους. Θα ασχοληθούμε με τη ΣΕΠΟΛ, με την Ευρωπόλ, με την Eurosur, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε όλες αυτές οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να ξεχνάμε το στρατηγικό ρόλο που διδραματίζουν οι ευρωπαϊκοί αυτοί οργανισμοί προκειμένου να καταφέρουν να συντονίσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διάφορα επίπεδα λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά συγκεκριμένα την Frontex, τι θα κάνουμε με τη Frontex, τι ελπίζουμε να πετύχουμε στα πλαίσια της Frontex Αν το ζήτημα των συνόρων αποτελέσει αποκτήσει μάλλον κεντρικό χαρακτήρα, όπως πραγματικά εμείς το επιθυμούμε, να αποκτήσει κεντρικό ρόλο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τότε ο οργανισμός ο οποίος θα πρέπει να ελοποιήσει όλα τα προγράμματά μας δεν μπορεί να είναι ένας μικρός οργανισμός με λίγα χρήματα, με ελάχιστους πόρους, Ξέρετε, το ζήτημα αυτό αφορά πάρα πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθότι είναι αρχή αρμόδια για τον προπολογισμό. Χρειαζόμαστε την απαραίτητη χρηματοδότηση και βελτίωση της Frontex, προκειμένου να μπορεί να ελοποιήσει τους στόχους και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης, η κυρία Σίπελ αλλά και άλλοι με ρώτησαν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να ελοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία ήδη ξεκίνησαν ως πρωτοβουλίες από τις προηγούμενες προεδρίες και να καταφέρουμε παράλληλα να συμπληρώσουμε ό,τι εκκρεμεί αυτή τη στιγμή με δικέ μα νέε πρωτοβουλίε. Και αναφέρομαι εδώ πέρα και στην κυρία Βίξτρομ, η οποία γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση, καθότι η εισηγήτρια για το ζήτημα των φοιτητών, των σπουδαστών που έρχονται από τρίτε χώρε. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ και θεωρώ και εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερη ελκυστική ήπειρο καθότι έχει έναν τεράστιο πλούτο πολιτισμικό και πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα τα ζήτημα της τρομοκρατίας, γνωρίζουμε προφανώς πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα λεπτό και ευαίσθητο ακριβώς επειδή εντάσσεται στο ζήτημα αυτό και το ζήτημα των μοναχικών αυτών λύκων, μεμονωμένων μαχητών, των ξένων μαχητών, οι νέε αυτέ μορφέ δηλαδή εγκληματικότητα που θέτουν κινδύνο την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε όλα αυτά τα προγράμματα αστυνομική συνεργασία αλλά και τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα δεδομένα PNR, τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα φύση e σύνορα, όλα αυτά δηλαδή τα προγράμματα τα οποία βοηθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσει καλύτερα πώς μπορεί να διαχειριστεί την ευκταία αυτή κινητικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε και με το πολύ λεπτό και ευαίσθητο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία επενδύει στα σύνορά τη δεν θα πρέπει να ενισχύει μόνο τι αρμόδιε υπηρεσίε τη, αλλά θα πρέπει να κάνει και κάποιε συγκεκριμένε νομοθετικέ επιλογέ που θα είναι σε θέση να προασπίσουν καλύτερα τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να είμαι σύντομο στην παρέμβασή μου και ήδη ο Πρόεδρο Μωράε, μόλον ότι δεν το βλέπετε αυτή τη στιγμή, μου λέει ότι θα πρέπει να ολοκληρώσω. Προσπάθησα λοιπόν να είμαι ευσύνοπτο στην παρέμβασή μου αυτή. Και πρέπει να σας πω και ολοκληρώνω ότι τίθεται πάντα και αυτό το ζήτημα των ανήλικων, το μη συνοδευόμενων ανήλικων, κάθε φορά που μιλάμε για μετανάστευση. Προφανώς και το ζήτημα αυτό αποτελεί ανθρωπιστική προτεραιότητα και θα πρέπει να επικεντρώνονται σε αυτούς οι ανθρωπιστικέ μα δράσει. Αναφερόμαστε κυρίως σε παιδιά ή εφήβους 17 ετών. Πολλές φορές όμως μιλάμε και για πραγματικά μικρά παιδιά. Αναφερόμαστε στους ασυνόδευτους ανήλικους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του ε, προβλήματος αυτού και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δείξουμε ότι είμαστε αντάξιος Ευρωπαίοι, ότι έχουμε πραγματικά δημιουργήσει εδώ πέρα την πιο σημαντική παγκόσμια δημοκρατία. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο το έργο που έχετε να απαντήσετε ε, συνολικά και εκτενώς, αλλά έχουμε άλλους 23 συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν και πρέπει να τελειώσουμε και στις 12.30. Ε, είναι λοιπόν τεράστιο το έργο σας και παρακαλώ τον κύριο Λάντο να απαντήσει και θα πρέπει να απαντήσετε και μετά. Λοιπόν, τώρα απαντήστε σύντομα, θα έχετε την ευκαιρία και στη συνέχεια. Έχετε και δευτερολογία. Ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε κάποιες απαντήσεις ε, στον τελευταίο γύρο απαντήσεων, αλλά θα ήθελα αυτή τη φορά να αναφερθώ περισσότερο στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς επίσης και στο ζήτημα της χρηματοδότησης της Eurojust. Καταλαβαίνετε, τα ζητήματα αυτά αποτελούν αρμοδιότητα τη δική σα επιτροπή. Όσον αφορά τι διαπραγματεύσει, ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι διαπραγματεύσει όσον αφορά δηλαδή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Συμβούλιο θα δει ποια θα είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ποιε σε ποιες συμπεράσματα θα καταλήξουν σχετικέ διαπραγματεύσει. Θεωρώ πραγματικά ότι είναι πολύ δύσκολο να λυθεί ο γόρδιο δεσμό που έχει προκύψει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον ρόλο που θα πρέπει να έχει αυτό το νέο θεσμικό όργανο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πρέπει να καταφέρουμε να δούμε ποιε θα είναι οι αρμοδιότητε τη αγγελία αυτή και πώ θα καταφέρουμε χρηματοδοτικά αλλά και μέσω προσωπικού να στηρίξουμε τη νέα αυτή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και σίγουρα το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δευτερεύον. Αλλά πρέπει πρώτα να επιληθεί το ζήτημα της θεσμικής αρχιτεκτονικής, αν θέλετε. Το ζήτημα της ε, οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων αυτής της αγγελίας. Όσον αφορά τώρα την ε, απόφαση και τις δικαστικές αποφάσεις για την συντήρηση διατήρηση των δεδομένων, υπάρχει πάλι μια σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία επεξεργάζεται το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι θέλει να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις πάρα πολύ σύντομα. Όσον αφορά πάλι το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συμφωνώ με την προσέγγιση που αναφέρθηκε από την κυρία Σίπελ. Επαναλαμβάνω ότι το σημείο έναρξης των διαπραγματεύσεων πρέπει προφανώς να είναι το ζήτημα της καταπολέμησης των, της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι γίνανε διάφορες προτάσεις για την αρμοδιότητα που θα πρέπει να έχει αυτή η εισαγγελιακή αρχή και πολλοί στη συνέχεια προσπάθησαν να διευρύνουν αυτή την αρχική αρμοδιότητα. Εγώ πάντως νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε ραλιστικοί θα πρέπει να επιμείνουμε ακριβώς σε αυτό το τομέα υπεράσπιση οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν μειώθηκε το πεδίο εφαρμογής της εισαγγελικής αυτής αρχής. Θα πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ενέχεται, καταλαβαίνετε, και ένας κίνδυνος κάθε φορά που διευρύνουμε τις αρμοδιότητες αυτές, αυτής της αγγελικής αρχής. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι κατά την εξέλιξη των πραγματεύσεων για το φάκελο αυτό είναι αναγκαίο από κοινού να δούμε πώς θα καταφέρει η Ευρωπαϊκή αυτή εισαγγελική αρχή να ενισχύσει περισσότερο τις δικονομικές εγγύησεις. Η Ιταλική λοιπόν Προεδρία θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το εξειδικευμένο αυτό ζήτημα. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του δικαιώματος λήθης, το Συμβούλιο είπε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως ε, η ε, οδηγία όσον αφορά τις μηχανές έρευνα στο διαδίκτυο. Θα λάβει υπόψη της λοιπόν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου η Ιταλική Προεδρία. Νομίζω πάντως ότι στη σχετική δικαστική απόφαση υπάρχουν ήδη κάποια στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε και σε μια κοινοτική νομοθεσία. Ήδη όμως είδαμε ότι στις διμερείς επαφές που είχαμε στο σχετικό συμβούλιο υπάρχει χάσμα απόψεων αυτή τη στιγμή, πολύ μεγάλη απόκληση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτος μας στόχος λοιπόν είναι να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή τοποθέτηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά πάντα το δικαίωμα της λήθης. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του εντάλματος σύλληψης, του διεθνούς εντάλματος σύλληψης, του ευρωπαϊκού με συγχωρείτε εντάλματος Ξέρετε ότι είχαμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα προϊόντος του χρόνου. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του εντάλματος σύλληψης, αλλά θα πρέπει στα πλαίσια του εντάλματος σύλληψης να προασπίσουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Όσον αφορά τώρα πάλι το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων. Αναφέρομαι εδώ πέρα στο ερώτημα της ε, κυρίας Έρνστα, Συντοπιώ ότι ε, συνειδητοποιώ την αγανάκτησή της. Πάντως εγώ επαναλαμβάνω την τοποθέτηση της Ιταλικής Προεδρίας. Εμείς προτιμήσαμε κανονισμό και όχι τόσο οδηγία και νομίζω ότι υπήρχαν οι κατάλληλοι λόγοι για να γίνει η επιλογή αυτή. Πρόθεση δηλαδή της λύσης του κανονισμού και νομίζω ότι και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει μια καλύτερη εναρμόνιση των κοινοτικών διατάξεων και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω κανονισμού στην συζήτηση που έγινε στο άτυπο Συμβούλιο του Μιλάνου φάνηκε ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών συμφωνεί με αυτή την επιλογή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική η προϋπόθεση αυτή, να έχουμε δηλαδή ένα κανονισμό, γιατί θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη δυνατή ομοιόμορφη υλοποίηση των διατάξεων σε κοινοτικό επίπεδο. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τώρα την οδηγία, όλες οι προηγούμενες προεδρίες, και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, αποφάσισαν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον κανονισμό και όχι τελικά στην οδηγία. Όλες οι προηγούμενες προεδρίες θεώρησαν ότι ο κανονισμός αποτελεί μια πολύ πιο αποτελεσματική λύση. Οι εργασίες λοιπόν οι για τον κανονισμό απαιτούν πολύ σκληρή εργασία από όλους μας. Καταλαβαίνετε ότι στον τομέα της δικαιοσύνης ο κανονισμός αυτός αποτελεί το πιο φιλόδοξο νομοθέτημα το οποίο είχαμε τελευταία χρόνια. Επίσης, ε, τα κράτη-μέλη, τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε για το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο προτού προχωρήσουμε σε επιμέρους λεπτομέρειες όσον αφορά δηλαδή τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία. Και νομίζω ότι η απέτηση αυτή είναι καθόλου λογική. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία προτιμούν την λύση της οδηγίας και αυτά αναφέρθηκαν σε κάποια προβλήματα που μπορούν να προκύψουν, πολιτικά προβλήματα σε σχέση με τις επιλογές που έχει κάνει στην πρότασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο όμως θα πρέπει να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση στα πλαίσια του Συμβουλίου δεν έγινε καμία συζήτηση προκειμένου να σταματήσουν οι εργασίες για την οδηγία. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε, να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Δεν έχουν προκύψει λοιπόν προβλήματα ούτε με τον κανονισμό ούτε με την οδηγία και δεν ισχύει αυτό το οποίο υπόθηκε από ορισμένου ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ζήτησαν στα πλαίσια του Συμβουλίου να σταματήσει οποιαδήποτε εργασία έχει να κάνει με την οδηγία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ένα ακόμα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Στη συνθήκη λέγεται ότι η πρωταρχική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων είναι και η πρόθεση και η προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια μόνο έρχεται το ζήτημα της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Ως προς αυτό λοιπόν, ως προς αυτό, λοιπόν θεωρώ ότι ομόφωνα στο Συμβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία να αναφερθώ και στα όσα είπε η κυρία Φεράρα. Δεν νομίζω ότι είναι επί του παρόντος ρεαλιστικό να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή η οποία θα ασχολείται με την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Νομίζω ότι είναι πιο ραλιστικό να ξεκινήσουμε την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εργασία που θα πρέπει εμείς να επιτελέσουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε το κατάλληλο αρχικό αν θέλετε πλαίσιο για τη σύσταση αυτού του οργανισμού είναι καταρχάς να πετύχουμε μια ομογενοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά τη δίμευση και την κατάσχεση. Και για τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο και να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις που προέρχονται από την προηγούμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΚΡΙΜ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όμω θα πρέπει να επιβαρύνουμε τη νέα εισαγγελική αρχή με μια τέτοια αρμοδιότητα. Δεν θα ήταν σωστό κάτι τέτοιο. Α έχουμε λοιπόν μια ρεαλιστική προσέγγιση για τη σύσταση αυτού του οργανισμού. Τέθηκε ένα ακόμα ερώτημα που έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένε Η Επιτροπή θα διεξάγει έναν γύρο διαπραγματεύσεων πριν το καλοκαίρι με τις Πολιτείες και έναν δεύτερο γύρο το Σεπτέμβριο. Μέχρι το φθινόπωρο νομίζω ότι θα έχουμε ήδη ένα κείμενο στα χέρια μας και θα μας σε θέση αυτή τη στιγμή να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων αυτών. Καταρχάς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στην προηγούμενη υπουργική διάσκεψη, οι Ηνωμένε Πολιτείε είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα δικαιοδοτικό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό αποτελεί σημαντικό το επίτευγμα γιατί για πρώτη φορά αποδέχθηκαν την υποχρέωση αυτή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Σας ευχαριστώ. Um, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε λίγο χρόνο πια στη διάθεσή μας. Θα τα καταφέρουμε μόνο αν όλοι περιοριστούν στο ένα λεπτό θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι αδύνατον. Αν το κάνετε όλοι, θα μπορέσουμε να ακούσουμε και τα συμπεράσματα των Υπουργών, οι οποίοι έδωσαν ολοκληρωμένες απαντήσεις. Οπότε περνάμε αμέσως στον κύριο Δίας Τεμέρα. Θα σηκώσω αυτό το γελίο αντικείμενο ε, για, στο ένα λεπτό. Αν θέλετε να είστε ευγενείς στους συναδέλφους σας, περιοριστείτε στο ένα λεπτό αν θέλετε αμέσως να γίνετε αντιπαθής ή μη δημοφιλής, να με απολύσετε την πρώτη μέρα που έχω αναλάβει είναι δικό σας θέμα. Λοιπόν, θα το χτυπήσω στο ένα λεπτό. Είναι εντυπωσιακό το ότι μπορεί κανείς να κάνει σε ένα λεπτό. Λοιπόν, κύριε Ντεμέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Για την Ευρωπόλ και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι κόκκινη γραμμή για μας αυτό. 610 βουλευτές με υποστηρίζουν. Δεν θέλουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που προτείνει η Ιταλική Προεδρία, ούτε εκείνον που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε θέλουμε εκτελεστική επιτροπή για να παίρνουν τρει άνθρωποι τι αποφάσει. Θέλουμε διοικητικό συμβούλιο για να λαμβάνονται από 23 για τη μετανάστευση. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τον όρο παράνομη μετανάστευση. Τι λέμε ε, παράτυπη ε, ή λάθρο μετανάστευση. Δεν τους λέμε παρανόμους. Τρίτον, για να προστατεύσουμε ε, την ελευθερία ε, διέλευσης θα πρέπει να προστατεύουμε τα εξωτερικά σύνορα που είναι και χερσαία από θάλασσα, ξηρά και αέρα δηλαδή και από ποτάμια. και υπάρχει ομοφωνία ε, για το ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, γιατί ξαφνικά στην Ελληνική Προεδρία 11 χώρε διαφωνούσαν. Ευχαριστώ. Η Σιλβί Γκυγιόμ, παρακαλώ. Ε, Προ την κατεύθυνση που ανέφεραν πολλοί από του συντονιστέ, κάποιε διευκρινήσει επιπλέον για την συνολική προσέγγιση στο θέμα των μετανάστευσης. Τι έγινε με το, στο προηγούμενο συμβούλιο. Υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις Άρα δεν ανταποκρίνονται στην πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουν. Πώς θα σκοπεύετε να δουλέψετε για την δική μας μεταναστευτική πολιτική που να είναι συνεπής και αποτελεσματική και τι προβλέπετε ε, να συνεργαστεί, στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη ώστε να φροντίσετε ότι το θέμα της μετανάστευσης θα αντιμετωπιστεί πιο ολοκληρωμένα. Τώρα για την ε, νόμιμη μετανάστευση. Θεωρείτε ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική νόμισης μετανάστευσης που να περιορίζεται στους, υψηλά, στους εργαζόμενους με τα υψηλά προσόντα και τέλος, όσον αφορά την κατανομή των ε, ευθυνών σε θέμα του ασύλου, αναφερθήκατε προηγουμένως στην πρόταση της Ιταλικής Προεδρίας για την αμοιβή αναγνώριση μεταξύ κρατών μελών της απόφασης ε, για το άσυλο, αλλά η οποία όμως ε, έφυγε από τις στρατηγικές αποφάσεις του Συμβουλίου. Ποια είναι η στρατηγική που σκοπεύετε να ακολουθήσετε για να προχωρήσουμε πέρα από τα λόγια για την ελληνική, για την ανάληψη των, ε, τους των ανθρώπων που κινδυνεύουν να πνιγούν. Μία πρόταση προς τους Υπουργούς, αν δεν έχετε αντιρρήσει. Αν υπάρχει κάποια σοβαρή ερώτηση την οποία δεν έχετε ε, χρόνο να απαντήσετε, μπορείτε να, να απαντήσετε και γραπτά εκ των υστέρων. Ε, πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Ε, τώρα, έχετε επόμενη ερώτηση. Η κυρία, η κυρία ε, Ιντοβέλ, αλλά Άννα έχει το λόγο πρώτο. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Ήμουν εισηγήτρια ε, για την οδηγία τότε. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να αντιμετωπιστεί η ζήτηση στις διακίνη, παράνομης διακίνηση ανθρώπων. Δεν έχετε μιλήσει στο πρόγραμμά σας για την αντιμετώπιση της ε, ζήτησης αυτή ε, αυξάνεται εντυπωσιακά στην Ευρώπη και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ζήτηση στα κράτη-μέλη. Το άρθρο 18 της οδηγίας αναφέρεται στη σημασία της αντιμετώπισης της ζήτησης και στο άρθρο 23 αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει το 2015 και 2016 να επενέλθουν στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή για να πούν πώς ακριβώς ε, κινηθήκαν για να αντιμετωπιστεί αυτή η ζήτηση σε σχέση με την οδηγία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρετε αυτό και είναι σαφές ότι τίποτα δεν υπάρχει στο πρόγραμμά σας. Τι σκοπεύετε για την, να, να, κάνετε για να αντιμετωπιστεί η ζήτηση. Επόμενη η Σόφη θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένη με το πώς προχωρούν τα πράγματα. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν μιλήσει 4-5 λεπτά, εδώ στο τέλος μας μένει ένα λεπτό, στο τέλος δεν θα πάρουμε απάντηση. Τελικά, τι σκοπεύει να κάνει η Ιταλική Προεδρία για να απελευθερώσει τις ε, διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό για τη διαφάνεια. Δεύτερον, η Ιταλική Προεδρία συμφωνεί ότι αποτελεί πραγματικό έσχος ο τρόπος με τον οποίο το Συμβούλιο προσπαθεί να παρακάμψει ε, το, την αίτηση για απόφαση του δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναφέρονται στα πρακτικά όταν έχουν θέση ή έχει σκοπό να το κάνει αυτό η Ιταλική Προεδρία εθελοντικά σε συνεργασία ίσως με άλλες χώρες που πιστεύουν όντως τη διαφάνεια. Δεύτερον, επί πέντε χρόνια παλεύω για να έχω πρόσβαση σε ένα έγγραφο και το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ μου στις 3 Ιουλίου. Πότε το Συμβούλιο θα ανταποκριθεί στο αίτημά μου επιτέλους και τέλος έχουν ε, υποβληθεί πολλές ερωτήσεις σχετικά με την ακύρωση της ε, ε, οδηγίας διατήρησης και δεν άκουσα. Πιστεύετε ότι είναι έσχος που δεν έχουν ανακληθεί οι, νομι... οι εθνικές νομοθεσίες και ίσως θα πρέπει να έχουμε κατεπίγουσα νομοθεσίες σε καιρό ειρήνης. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που σκοπεύετε να έχετε κοινή συνεδρίαση με τους Υπουργούς Εξωτερικών, γιατί πράγματι πολλά ε, από τα προβλήματα έχουν σχέση. Η Λιβύη δεν είναι χώρα που υπάρχει αστάθεια, είναι ένα αποτυχημένο κράτος γιατί η Ευρώπη εν μέρει αποφάσισε, δεν κατάφερε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει προτείνω στη συνεδρίαση αυτή να επικεντρωθείτε στον τρόπο με τον οποίο ε, ε, σπαταλώνται οι πόροι του ναυτικού για να ε, μην και δεν είναι αποτελεσματική η δράση της ΕΠΑ. Επίσης, υπάρχει και η νόμιμη μετανάστευση. Τώρα, το θέμα της αναθεώρησης της οδηγίας για το ξέπλυμα ε, χρήματος. Πού βρισκόσαστε και θα επιδιώξετε να συμπεριληφθούν και τα εθνικά μητρώα των υπευθύνων των εταιριών έτσι ώστε να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της ε, απάτης στο επίπεδο των φόρων, στο επίπεδο της απόκρυψης εσόδων και τις εγκληματικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Η Σεσίλ. Grazie. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους Υπουργούς. Θα θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα. Πρώτον, στην Ιταλία, προφανώς έχουμε τη σημαντικότητα αυτή Προεδρία αυτή τη στιγμή, πώς θα καταφέρουμε να προωθήσουμε την καταπολέμηση της παρίσφρησης εγκληματικών οργανώσεων στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα καταφέρουμε επίσης να καταπολεμήσουμε την αδιαφάνεια και οποιαδήποτε διαφθορά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έπειτα έχουμε το ζήτημα του hate speech, της βίας που εκδηλώνεται μέσω δηλώσεων μίσους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της Ιταλικής Προεδρίας για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Το ζήτημα επίσης της υπηκότητας, της ηθαγένειας, ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ιταλία ιδιαίτερα διότι θα πρέπει να υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινά κριτήρια όσον αφορά το ζήτημα αυτό της υπηκότητας. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να δεσμευτεί περισσότερο η Ιταλία για το ζήτημα της καταχώρησης των παιδιών εκείνων από γονείς οι οποίοι δεν έχουν έγγραφα ταυτοποίηση στην δαφική επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χον Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ, ευχαριστώ Κλοντ. Εδώ είμαι. Θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ ότι καλύτερο στην Ιταλική Προεδρία και χαιρετίζω και τους υπουργού και είχα την ευκαιρία και στο παρελθόν με τις προηγούμενες ιδιότητες του Προέδρου εδώ της Επιτροπής και Υπουργού Δικαιοσύνης της Ισπανίας να συνεργαστώ. Αναφέρθηκε στα εγκλήματα μίσους ο κύριος Αλφάνο. Το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο από το διεθνή του χαρακτήρα και από το γεγονό ότι εδράζεται ε, στις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική ε, πρωτοβουλία μετά από όθηση και του Συμβουλίου για μια νέα νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους. Επίσης, πολύ σημαντικά για το χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης είναι δύο θέματα όπου το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν συμφώνησαν αλλά το Συμβούλιο όχι για την προστασία των δεδομένων. Ποια είναι η ρεαλιστική προοπτική προόδου που θα μπορούσε να αφορά το εξάμεινο της Ιταλίας και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ ξέρετε είμαι εισηγητής ε, το θέμα τους για την προστασία και την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και δηλώνω προθυμία για τον τριμερή διάλογο όσο γίνεται να συνεισφέρω στην αποτελεσματική και γρήγορη λειτουργία. Αυτό το θέμα είναι ε, ο προάγγελος οι ε, ε, εισαγγελία θα πρέπει να εγκριθεί κατά τη διάρκεια του δικού σας εξαμήνου. Ευχαριστώ πολύ Χουάν. Η Τζιν Λάμπερτ. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ερώτηση που αφορά σε αυτό που λέγαμε για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, ένα από τα οποία προφανώς είναι η συμμεταχείριση και η αποφυγή των διακρίσεων. Να πούμε δύο λόγια περισσότερο, αν είναι δυνατόν, για το πώς βλέπετε τις προσπάθειες για την καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Φερρυπίν, αντιμετώπιση, ε, ποιότητα αντιμετώπισης με βάση την φιλετική εθνική προέλευση και γενικότερη στρατηγική και επίσης το θέμα της Παράταση της νομοθεσίας ε, κατά των διακρίσεων γιατί υπάρχει μια νομοθεσία η οποία έχει μείνει εκεί στο ράφι να δούμε τι θα γίνει επ' αυτού. Ε, και βεβαίως ο εισηγητής του Κοινοβουλίου θα είναι πρόθυμος να βοηθήσει το Συμβούλιο αν χρειαστεί. Αλλά αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα τα, επί των οποίων πρέπει αυτή τη στιγμή κάτι να κάνουμε. Επόμενος, κυρία Τάλι Βέριαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, απευθύνω την ερώτησή μου στον κύριο Αλφάνο και αφορά για την, την επιχείρηση Μάρεν Όστρομ. Ξέρουμε ότι διασώζονται εκατοντάδες άνθρωποι από τη Μάλτα, ένα μικρό νησί της Μεσογείου, γνωρίζω ότι πρόκειται για μια εκτεταμένη επιχείρηση που ασκεί πίεση στους πόρους της χώρας μας. Γνωρίζουμε ότι η Ιταλία θέλει να εμπλακεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχείρηση αυτή. Οπότε ρωτώ, τι ακριβώς περιμένει η Ιταλία. Δηλαδή περιμένει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την επιχείρηση, τη Μαρενόστρουμ, ή περιμένετε οικονομική βοήθεια και θεωρείται ότι η Ιταλία πληρώνει, αν λάβουμε υπόψη μας ότι 9 εκατομμύρια ευρώ το μήνα πληρώνει η Ιταλία από αυτού. Τι περιμένει η Ιταλία και ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής που έχετε κατά νου. Ευχαριστώ. Η επόμενη κυρία Περί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επανειλημμένα ακούστηκε ότι οι τζιχαντιστές που πάνε στη Συρία και στο Ιράκ και συνέχεια επιστρέφουν είναι Ευρωπαίοι. Και θέλω να ρωτήσω, τι προτίθεται να κάνει η Ιταλική Προεδρία για να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρούν ότι οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών συνεργάζονται με βέλτιστο τρόπο για να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους μαχητές του τζιχάτ και πώς θα βελτιωθεί η συνεργασία όταν πρόκειται στην πρόληψη ε, για να μην υπάρχει αυτή η ε, ακραία εμφάνιση ε, και η κλιμάκωση. Ευχαριστώ.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 ακούστηκε επανειλημμένος από την εποχή που ξεκίνησε η κρίση στη Μεσόγειο και στη συνεδριά της Επιτροπής ότι μπορεί η παράνομη μετανάστευση να σταματήσει με το να ανοίξουν νέοι δρόμοι εισόδου στην Ευρώπη. Αυτή όμως η προσέγγιση δεν μου φαίνεται ότι θίγει το βασικό πρόβλημα, δηλαδή ότι σήμερα όπως είναι η Ευρώπη δεν μπορεί να προσφέρει απασχόληση στις εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που είναι ανειδίκευτοι, ούτε μπορεί οικονομικά και κοινωνικά να αντέξει έναν μη ενταγμένο μεταναστευτικό πληθυσμό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τώρα η Ευρώπη έχει πετύχει στις προσπάθειες ένταξης. Τα προβλήματα παραμένουν ασχέτως από το αν οι άνθρωποι φτάνουν νόμιμα ή παράνομα στην Ευρώπη. Άρα θα ήθελα με δύο λόγια να ακούσω το στρατηγική σας προσέγγιση στο θέμα της αντιμετώπισης της μεταναστευτικής πίεσης χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο ούτε τα δικαιώματα αυτών που έχουν δικαίωμα προστασίας, ούτε τη συνοχή της κοινωνίας μας και τα θεμέλια των συστημάτων πρόνοιας που διαθέτουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Φόρκ Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βος. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη μαζική παρακολούθηση, όπως τα λέει και η έκθεση NSA. Και υπάρχει και το δικαίωμα στη λύθη που αναφέρθηκε. Έχω την αίσθηση ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα πλαίσιο για να μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το δικαίωμα στη λύθη και άλλα ε, πράγματα να μπορούν να τα διατηρήσουν. Τώρα, κατά πολέμηση της εγκληματικότητας ε, στο διαδίκτυο. Ε, ε, σχέση με την απόφαση του ΔΕΚ για την προληπτική διατήρηση και αποθήκευση δεδομένων. Πώς θα λυθούν τα προβλήματα. Αναφέρθηκε ο θρησκευτικός ε, φοντομεταλλισμός. Πρόκειται για τις αντοχές της ελευθερίας και των δικαιωμάτων μας που δοκιμάζονται και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, χρειάζεται και ένα δικονομικό ε, δίκαιο, σε περίπτωση δηλαδή που ε, συσταθεί. Ακριβώς το λεπτό επάνω τελείωσης. Η κυρία Μουσολίνη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ορλάντο στην παρέμβασή του δεν αναφέρθηκε στην πολιτική ευθύνη των δικαστών. Εμείς έχουμε πάρα πολλές εκκρεμούσες διαδικασίες κατά της Ιταλίας συγκεκριμένα και ενδεχομένως να προκύψουν κάποια προβλήματα. Δεν υπάρχει πλέον στην Ιταλία η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και δικαστικού συστήματος. Ας προσέξουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τα σοφρονιστικά ιδρύματα και τις φυλακές, μην ξεχνάτε ότι και εκεί πολλές φορές υπάρχει απαξιωτική αντιμετώπιση των παιδιών αλλά και των γυναικών, των μητερών τους. Ελπίζω και απευθύνομαι τώρα στον Υπουργό Αλφάνο ότι θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταποτελεμήσουμε διάφορα προβλήματα όπως τρομοκρατία ή παράνομη μετανάστευση. Αναφερθήκατε εσεί στην Frontex για την έντρα που θα μπορούσε να έχει στην Ιταλία ή ενδεχομένως να έχουμε ακόμα και έναν Ιταλό επικεφαλής της Frontex. Ως προς αυτό θα ήθελα να γνωρίζω πώς ακριβώς θα απορροφηθεί η επιχείρηση Mare Nostrum από τη Frontex. Τι θα γίνει επίσης με το Eurosur, το Ευρωπαϊκό Αυτοσύστημα Επιτήρησης των Συνόρων, που είχε ένα κόστος μέχρι πρόσφατα 338,7 εκατομμύρια ευρώ. Διόλου αμεληταίο το ποσό αυτό. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι ξένοι οι οποίοι φτάνουν στην Ιταλία και δυστυχώς ε, τη στιγμή πατάνε στο Ιταλικό έδαφος αντιμετωπίζονται απλώς σαν ένα νούμερο και όχι σαν άνθρωποι. Είναι πολύ, σημαντικό, είναι με συγχωρείτε λοιπόν να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε και για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Σφοντάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα και στους δύο Υπουργούς. Μια ερώτηση για τον κύριο Αλφάνο όσον αφορά την επιχείρηση Mare Nostrum. Σαφώς από τη μία πλευρά θα πρέπει να προστατεύσουμε όλα αυτά τα άτομα τα οποία έρχονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να αποφύγουν κάποια πολιτικά καθεστώτα, από την άλλη όμως θα πρέπει να διχειριστούμε και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άτομα αυτά τα οποία καταφθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τελευταίες αυτές μέρες είναι πάρα πολύ όπως βλέπουμε, τα άτομα αυτά τη στιγμή που δεν έχουν ταυτότητες, πώς ακριβώς θα ταυτοποιούνται, ποια διαδικασία εξακρίβωσης προβλέπεται, θα χρησιμοποιηθούν κάποια άλλα πιστοποιητικά, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έστω και πολύπλοκη διαδικασία εξακρίβωσης. Αυτή τη στιγμή επίσης τα άτομα αυτά ταυτοποιηθούν. Από τα άτομα αυτά πόσα τελικά θα έχουν το δικαίωμα αίτηση ασύλου. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία τελικά δεν καταχωρούνται σε κανένα μητρό και τελικά μπαίνουν περισσότερο στο περιβάλλον αυτό στο χώρο της παράνομης μετανάστευσης. Στη συνέχεια, τι κάνουμε με αυτούς τους παράνομους μετανάστες, πώς μπορούμε να τους διαχειριστούμε, τι κάνει η Ιταλική κυβέρνηση για παράδειγμα και πώς μπορεί να συνεργαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Ξέρετε ότι ιδίω σε περιόδους έντονης μεταναστευτική πίεσης ενδεχομένως να μην κάνουμε τίποτα με τα άτομα αυτά και ενδεχομένως να τίθεται τελικά να αμφιβόλω και η ίδια η διασφάλιση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Στη συνέχεια, ο κύριος Νάγκη. Α, είναι εδώ ο κύριο Σολτ, δεν σα είχα δει. Ζητώ συγγνώμη. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Αρφάνο, Σέγγεν, Ρουμάνια. Ρουμανία. Γιατί όχι. Δεύτερη ερώτηση. Κύριε Ορλάντο, αναφερθήκατε τα δικαιώματα. Αν ξέρατε τι γίνεται στην Ελλάδα, Σλοβακία και Ρουμανία, πώς μπορεί να βοηθήσετε τα κράτη-μέλη να ε, βοηθήσετε να στηρίξουν τα δικαιώματα των πολιτών τους. Κύριος Νάκη, είναι ή δεν είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούγεται, να θεωρείτε ότι είμαι ανακουφισμένος όταν κάποιος δεν είναι εδώ. Κύριε Νάγκη, έχετε το λόγο. Δύο πρακτικά ερωτήματα στον κύριο Αρφάνο που αφορούν τη μετανάστευση. Σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία. Ως Ευρωβουλευτής από την Σλοβακία, που είμαστε γείτονες της Ουκρανίας, εκατοντάδες χιλιάδες ε, μετανάστες για ανθρωπιστικούς λόγους μπορούν να εμφανιστούν στα σύνορά μας. Πρέπει να ε, είναι ενήμεροι για το τι ε, τους περιμένει. Δεύτερον, παράνομη οικονομική μετανάστευση. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Η πρόληψη αποτελεί μήπως πιθανή, τρόπο, πιθανό τρόπο αντιμετώπισης. Κυρίως στο, επειδή στο πλαίσιο της παράνομης εκείνης ανθρώπων οι άνθρωποι ακούν να τους υπόσχονται τη γη που ρέει μέντλι και γάλα και τελικά βεβαίως ε, δεν συμβαίνει αυτό. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα εξηγώντα στους ανθρώπους ότι οι παράνομοι μετανάστες δεν μπορούν να περιμένουν ότι θα στεγαστούν ε, δωρεάν και ότι, δεν θα, ε, ότι θα βρουν δουλειά επιπληρωμή και ότι αυτό ίσως είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε τους λαθροδιακινητές. Επίσης θυμάμαι ότι στο παρελθόν πριν πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα δεν είχαμε ε, σωστή ενημέρωση και ενδεχομένως μπορεί ακόμα να ισχύει αυτό, ακόμα και στην εποχή του διαδικτύου. Ε... Στη συνέχεια η κυρία Γκαβριέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αλφάνο επιμείνατε πάρα πολύ στην ενίσχυση ε, της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Τι σημαίνει αυτό, πολιτικές δηλαδή, όμως που μας δίνουν την αίσθηση ότι έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών. Ερώτηση. Βουλγαρία και Ρουμανία και χώρο Σέγγεν. Πότε θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Δεύτερον, θεώρηση διαβατηρίων με Ηνωμένε Πολιτείες και Καναδά. Έχουμε δύο χώρες στην Ευρώπη για τις οποίες δεν ισχύει και δεν γίνεται σεβαστή η αρχή της αμοιβαιότητας που μας είναι τόσο προσφυλής εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλά χάρη στην πρώην θητεία και το συνάδελφο Δίας Δεμέρα τον Οκτώβριο θα μας δώσουν μια συλλογική απάντηση. Πώς θα δεσμευτεί να προωθήσει αυτό το θέμα η Προεδρία σας. Κύριε Ορλάντο, η διακίνηση ανθρώπων, τι γίνεται με την οδηγία του Απριλίου 2011, τι κάνετε για να μπορέσουν όλες οι χώρες να τη μεταφέρουν στην ομοθεσία τους. Και ένα σημαντικό στοιχείο θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, την προσοχή μας για τη στρατολόγηση των θυμάτων με τα κοινωνικά δίκτυα και το ίντερνετ. Ε, Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Γιούρεκ. Ναι, ε, ευχαριστώ πολύ. Δύο εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες πέρυσι υπέγραψαν μία αναφορά και οι περισσότεροι αυτών ήταν Ιταλοί, ε, των υπογραφών δηλαδή. Και ερωτώ και τους δύο υπουργούς. Θα πρέπει και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών να την να τις δώσει συνέχεια. Πρόκειται για τη μη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, των αμβλώσεων ε, που μας απασχολεί. Θέλουμε να έχουμε ως αξίες ε, την αλληλεγγύη, ε, τη συνεργασία και να μην χρηματοδοτούμε τις αμβλώσεις. Αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ε, προσέκρουσε στην περιφρόνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την αγνόησε. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και είναι δύο εκατομμύρια Ευρωπαίοι που μάζεψαν υπογραφές. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, κυρία Σπινέλη. δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. για τις ε, δύο νέες αυτές μορφές Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι νέες θέσεις που μπορούμε να έχουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιο πρόγραμμα μπορούμε αυτή τη στιγμή να προωθήσουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Frontex, καθώς επίσης και τη δημιουργία κάποιων προστατευμένων ανθρωπιστικών οδών. Δεύτερο ερώτημα. Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Ερώτηση που απευθύνω προς τον Υπουργό Ορλάντο. Πώς είναι ποτέ ρεαλιστικό να συμπεριλάβουμε κάποια στιγμή στο μέλλον τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κρίμ και την καταπολέμηση της μαφίας και της απάτης, όταν από την άλλη θέλουμε να ασχοληθούμε τελικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία σαφώς έχουν παρισφρήσει και μαφιώσικες και κλιματικές οργανώσεις. Ε, Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αναφέρατε ότι θα κάνετε μια προσπάθεια για κοινή πολιτική ασύλου, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το σκέφτεστε αυτό? Ποιος θα αποφασίζει, δηλαδή, πόσους θα δέχεται κάθε χώρα. Αυτό είναι θέμα κάθε χώρας μόνης να το αποφασίζει. Για το πώς θα υποδεχθεί και ποιους θα υποδεχθεί τους ε, πρόσφυγες, τους μετανάστες, με έναν τρόπο αξιοπρεπή. Εγώ δεν είμαι καθόλου υπέρ μιας κοινή πολιτικής ε, ασύλου. Έρχομαι όμως ξανά σε αυτό που είπε ο κύριος Αλφάνο για τα χρήματα που θα δοθούν και πώς θα δοθούν έτσι ώστε να πιάσουν τόπο. Ε, πολύ καλό είναι αυτό, ωραία το λέτε. Εγώ προέρχομαι από μια βορειοευρωπαϊκή χώρα, τη Σουηδία, που ε, δέχεται δωδεκαπλάσιο αριθμό μεταναστών και τους υποδέχεται από άλλες ε, χώρες. Και ε, προφανώς έχουμε ε, χώρο να τους δεχθούμε, αλλά δεν μπορούμε στο δίνεκές να το κάνουμε αυτό. Ο Πρόεδρος. Παρακαλώ τους διερμηνείς να μας δώσουν λίγο περισσότερο χρόνο, να μην διακοπεί η συνεδρία και ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ να μας συμπαθάτε. Προφανώς δεν θέλω να φαίνω σε αυτή τη θέση και τους ομιλητές να πρέπει να απαντήσουν 24-25 ερωτήσεις. Ε, αυτά είναι ανέφικτα πράγματα. Σε, ούτε εσά για ερωτήσει ενό λεπτού. Σε κάποιε περιπτώσει βέβαια μπορεί να μην είναι και τόσο κακό αυτό. Να κάνετε ερωτήσει ενό λεπτού. Um, Αλλά νομίζω ότι θα βρούμε ένα καλύτερο τρόπο θα έπρεπε να το είχα προβλέψει αυτό. Είναι πολύ δραστήρια η Προεδρία. Καλύψατε όλα τα θέματα και έπρεπε να το είχα φανταστεί ότι θα είχατε γεννήσει τέτοιο ενδιαφέρον. Θα συζητήσω με τους συντονιστές ένα καλύτερο τρόπο συντονισμού για να έχουν την ευκαιρία τα μέλη και ιδιαίτερα τα νέα μέλη της Επιτροπής να πούν την γνώμη τους. Βεβαίως όλοι για τα ίδια θέματα μιλούν, αλλά ο καθένας να το δει από τη δική του σκοπιά και ως πολιτικός πάντα θες να λες τα ίδια πράγματα με τον προηγούμενο και να τα επαναλαμβάνεις για να εκλαμβάνεται αυτός πολιτική δήλωση. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τους δύο υπουργού αν έχουν την καλοσύνη για κάποιες ειδικέ απαντήσεις να τη στείλουν γραπτό αν γίνεται, να μην απαντήσετε τώρα. Απλώς να κάνετε μια τελική έτσι, καταληκτική τοποθέτηση ε, για να κλείσετε. Ευχαριστώ τους διερμηνείς για το χρόνο που μας δίνουν και για την υπομονή τους. Ποιος αρχίσει, ο κύριος Αραφάνο, παρακαλώ. Just, just one. If you can do what, this, what our speakers have done, maybe one minute. Ίσως ένα λεπτό, ένα ενάμιση, όπως και ο μιλητές μας, γιατί όχι. Για προσπαθήστε κι εσείς. Για να, να μην ειλικρινείς, κανείς δεν μίλησε ένα λεπτό. Μόνο βός, νομίζω. άλλη ένα ενάμιση. No, sarò davvero breve. Θα προσπαθήσω πραγματικά να είμαι πάρα πάρα πολύ σύντομος. Ε, μπορούν να είναι λακωνικοί ακόμα και οι Ιταλοί, λέει ο πρόεδρο. Ενδεχομένω δύο λεπτά τότε. Τρία, εντάξει. Όχι τρία. Δύο, δύο, δύο. Σα λέω δύο λεπτά μόνο. Μάλιστα. Στον τελευταίο αυτό γύρο ερωτήσεων είδαμε ότι υπάρχουν τα σημαντικά αυτά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μετανάστευση, εσωτερική ασφάλεια, τρομοκρατία θα πρέπει να καταφέρουμε να υποδεχθούμε προφανώς τους μετανάστες, αλλά παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Η στρατηγική λοιπόν που θα ακολουθήσουμε είναι ακριβώς αυτή. Να ενισχύσουμε δηλαδή τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να γίνει ένας πραγματικός παράγοντας εξωτερικής πολιτικής, Εκεί πραγματικά έγκυται, αν θέλετε, η λύση στο ακαθόδε ζήτημα της μετανάστευσης. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε την κατάλληλη διάκριση ανάμεσα στη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Θα το καταφέρουμε αυτό μόνο αν καταφέρουμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε εξωτερικό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας, μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πλέον τη δυνατότητα να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα ασφαλή χώρο στον οποίο μπορούν ειρηνικά να διαμένουν. Μας είπανε πολλοί συνάδελφοι ότι ε, ενδεχομένως να μπορούσαμε να προβλέψουμε και μια κάποια ενδυνάμωση οργανώσεων, οργανισμών όπως η Ευρωπόλ, η Eurosur, η ΣΕΠΟΛ, ως προς αυτό το αίτημα εγώ θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση η Ευρώπη δεν μπορεί να διατρέξει τον κίνδυνο να μην ολοκληρώσει το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε με τη Στοκχόλμη. Δηλαδή, στη Στοκχόλμη είχαμε συγκεκριμένε κατευθυντήρε γραμμέ, οι οποίε απέτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση ιδιαίτερα φιλόδοξα. Μετά το πέρα τη πενταετία του προγράμματο Στοκχόλμη, έχουμε πλέον εμεί ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να καταφέρουμε να ελοποιήσουμε μέσω τη απαραίτητη αναθεώρηση και επικαιροποίηση του στόχου που έχει θέσει το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. Είναι πολύ σημαντικό στο χώρο τη δικαιοσύνη και τη ασφάλεια Εξωτερικών Υποθέσεων να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα εκκρεμή ζητήματα. Να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την απόκληση απόψεων που εμφανίζεται πολλέ φορέ μεταξύ κρατών μελών. Με άλλα λόγια, να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε, αν θέλετε, τον εθνικό εγωισμό, το αποκαλέσω έτσι, που προβάλλεται από ορισμένα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή την ευρεία κοινοτική αρχιτεκτονική και να καταφέρουμε τελικά να ολοκληρώσουμε αυτό που κάποτε αποκαλούσαμε πρώτο πυλώνα. Να έχουμε από τη μια δηλαδή προστασία προστασία των δικαιωμάτων και από την άλλη μία προάσπιση δικαιωμάτων η οποία όμως να βασίζεται και στο σημαντικότατο ζήτημα της ασφάλειας. Το ζήτημα της μετανάστευσης, το είπα και το ξαναλέω, θα καθορίσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη όμως θα πρέπει να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και μια άλλη πρόκληση. Να γίνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση παράγοντας προσέλκυσης σημαντικών εγκεφάλων, επαγγελματιών ουσιαστικά παράγοντας νόμιμης μετανάστευσης προς την υπηρό μας. Νομίζω ότι όλες οι παρεμβάσεις που γίνανε σε αυτό το τελευταίο γύρο ερωτήσεων πραγματικά αναφέρθηκαν σε αυτή τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι με τη δική σας την Επιτροπή θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία όπως είχαμε μέχρι στιγμής και με τις υπόλοιπες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι, όπως σας είπα, στην πλήρη διαθεσή σας, προκειμένου να επιστρέψω εδώ στην Επιτροπή σας όποτε επιθυμείτε, προκειμένου να σας παρουσιάσω κάθε φορά πώς προχωρεί το σημαντικό το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ευχαριστούμε πολύ, Αντζελίνο. Ο Αντρέα έχει το λόγο. Όσον αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, εμείς ε, θεωρούμε ότι ε, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα πολιτικής φύσης και προφανώς μέσω ενός ρυθμιστικού πλησίου θα πρέπει να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό ενιαίο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία έχουν ήδη δημιουργήσει ένα καθεστώς προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών τους, αλλά πάλι όχι. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό προφανώς να εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου για το δικαίωμα λήθης. Θα συνεχίσουμε την πολύ σημαντική εργασία που ξεκίνησε η ελληνική προεδρία και εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παρακάμψουμε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσθέσω επίσης ότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει ο φάκελος αυτός κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας και μάλιστα ετέθηκε στη μερίσια διάταξη της άτυπης συνόδου, όπως σας είπα. Έχουμε αντιμετωπίσει όμως και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί έχει να κάνει με τη μεταχείριση των δεδομένων που διαθέτουν οι εθνικές αρχές, οι εθνικές δημόσιες αρχές. Δεν θεωρώ όμω ότι έχει γίνει ακόμα ό,τι είναι αναγκαίο και ότι πρέπει να γίνει. Αντίθετα θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να προχωρήσει περισσότερο ο φάκελος αυτός. Θα πρέπει λοιπόν οποιαδήποτε θετική πρωτοβουλία να την υποδεχτούμε. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλλον συγγνώμη την απόφαση της, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας πω το εξής. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται κάποια ομοφωνία στο Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση δεν είπα ότι υπάρχει ομοφωνία. Είναι σημαντικό όμως να καταφέρουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνένεση. Και η συνένεση αυτή μεταξύ κρατών μελών σε καμία περίπτωση θα πρέπει να βάλει κατά των ίδιων των θεσμικών οργάνων. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε τελικά σε ένα απλό συντονισμό των εθνικών δικαιοδοσιών που δεν θα μας επιτρέπει τελικά να δρούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να δρούμε αυτόνομα. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να πετύχουμε αυτή την κατάλληλη ισορροπία. Έχουμε ήδη επιδείξει όμως ένα συλλογικό πνεύμα, θα πρέπει να πετύχουμε μέσω της συλλογικότητα την κατάλληλη ισορροπία. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε όμως τόσο πολύ το συμβασμό ώστε να καταλήξουμε τελικά με μια συνεντική μεν απόφαση η οποία θα είναι άνευ νοήματος και που τελικά θα βάλει κατά της του ίδιου του οργάνου αυτού που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Τώρα, η απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν γίνεται βέβαια η απάτη αυτή από την μαφία, τότε προφανώς και η μαφία θα αποτελέσει τμήμα της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη στιγμή όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να οριοθετήσουμε ακριβώς αρμοδιότητες. Και είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να επιβαρύνουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή με κάτι το οποίο μοιάζει με το δικό μας το Ιταλικό άρθρο 416α. Πάντως έχουν ε, σημαντηθεί, θα πρέπει μάλλον να σημειωθούν, ε, να πρέπει να σημειωθεί πρόοδος και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Όπως σας είπα, στο ζήτημα της κατάσχεσης και της δίμευσης. Υπάρχει μια κάποια οριμότητα για το ζήτημα αυτό. Έχουμε καταβάλει προσπάθειες και νομίζω ότι μπορούμε κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας να επιτύχουμε σημαντικότερη πρόοδο όσον αφορά τη συμπερίληψη των δύο αυτών ζητημάτων κατάσχεση και δίμευση στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε προσεκτικά αυτά που είπατε. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία μαζί σας για την εσωτερική ε, στρατηγική ασφάλειας, εσωτερικής ασφάλειας 2014-2020 και ε, προσβλέπουμε και στην αξιολόγηση της οδηγίας για την Μεσόγειο και για την ε, δικαστική συνεργασία για όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας μέχρι στιγμής και εκτιμούμε πάρα πολύ την παρουσία σας και την παρουσία σας. Ευχαριστώ και τα μέλη.